matter. Because if I speak and they enter, then somebody has to make I them do sit it down. Okay. Uh, Dear colleagues, I would like to start the meeting uh, with the announcement of the decisions made at the level of coordinators. Uh, we Να ξεκινήσω με τι ανακοινώσει που προέκυψαν από την συνάντηση των συντονιστών σήμερα το πρωί. Καταρχήν να σα ενημερώσω ότι η συζήτηση τη γνωμοδότησης ΑΦΚΟ για την TTIP την Διατλαντική Συμφωνία ε, ε, αναβλήθηκε μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας. Ε, θα γίνει ε, ανταλλαγή απόψεων στις 6 Φεβρουαρίου, μετά τροπολογίες μέχρι τις 2 Μαρτίου και στις 17 ε, Μαρτίου θα, θα ψηφιστεί στην ΑΦΚΟ, στην Επιτροπή σταματικών Υποθέσεων εδώ. Όποιοι έχετε σοβαρές τροπολογίες Παρακαλώ να έρθετε σε επαφή με τον εισηγητή για να προετοιμαστείτε πριν τη συνεδρίαση. Έχουμε διερμηνία και στα λετωνικά, να σας το πω και αυτό. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την ε, αποστολή στη Ρήγα των συντονιστών, ε, ή μάλλον οι συντονιστές συμφώνησαν ε, να γίνει μεταξύ της 18 και της 20 Μαΐ, Μαρτίου αυτή, ε, αυτή η επίσκεψη. Συμφωνήσαμε επί της αρχής να κατανεμηθούν οι θέσεις ε, σύμφωνα με τον κανόνα don't, αλλά επιετήσιας βάσεως. Έτσι, για όλες τις ε, ε αποστολές επισκέψεις μαζί και μετά η κάθε μία πολιτική ομάδα ε, αν επιθυμεί και σε συμφωνία με μια άλλη πολιτική ομάδα μπορεί να κάνει ανταλλαγή θέσεων. Αλλά ο συνολικός αριθμός θέσεων για κάθε ομάδα θα καθοριστεί με τον νόμο του DONT συνολικά επί της βάσεως. Οι πολιτικές ομάδες ε, πρέπει να ενημερώσουν τη γραμματεία για το ποιοι είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν στην ε, επίσκεψη στη Ρήγα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Έξι θέσεις ...συν θέση της Πρόεδρου. Επίσης, πρότεινα και συμφωνήσαμε να διοργανωθεί μια διακοινοβουλευτική συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια μετά το καλοκαίρι, μάλλον τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, θα το αποφασίσουμε. Ζητήσαμε από τις πολιτικές ομάδες να μας υποβάλουν προτάσεις για θέματα ε, για αυτή την συνάντηση και ε, το νωρίτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Επίσης, ζητήθηκε να ερμηνεύσουμε τους ε, διαδικαστικούς κανόνες σε ό,τι για ένα θέμα που έχει σχέση με την δήλωση οικονομικών συμφερόντων από πλευρά των Επιτρόπων πριν τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Αποφασίσαμε το αίτημα αυτό να το προωθήσουμε στην ομάδα εργασίας που έχουμε δημιουργήσει για την αναθεώρηση των, ε, του, των, διαδικαστικών κανόνων ε, προκειμένου να απαντήσει. Αυτά. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ε, Η κυρία Λουκασέβιτσα, εκ μέρους της Λετωνικής Προεδρίας, θα μας παρουσιάσει ε, το πρόγραμμα της Λετωνικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά τις δικές μας ε, αρμοδιότητες. Εκτός και αν θέλει και να υπερβεί τις αρμοδιότητες μας στα θέματά μας και να μας παρουσιάσει και τις υπόλοιπε προτεραιότητες. Uh, uh, Ευχαριστώ κυρία Χίμπνερ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ε, είναι μεγάλη χαρά που είμαι παρούσα εδώ να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας και να συζητήσω λεπτομεριακά τα σημαντικά θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής σας. Πριν παρουσιάσω τις προτεραιότητες, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διασφάλισε μια ομαλή θεσμική μετάβαση αυτό σημαίνει ότι η Προεδρία μας ε, ξεκινάει σε ένα νέο θεσμικό κύκλο. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να δώσουμε νέα όθηση στην εργασία της Ένωσης για να έχουμε αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κόσμος ε, σημειώνει δυναμικές ε, οικονομικές από πλευράς ασφαλείας και γεωπολιτικές αλλαγές και προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί. Οι συνθήκες μας δίνουν ε, ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για να το πράξουμε, αλλά από εμά εξαρτάται να δράσουμε, να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και να περιφρορίσουμε τις αξίες μας. Μια τέτοια πρόκληση δυστυχώς ε, κατέστη απόλυτα σαφής στις 7 Ιανουαρίου μέσω των ε, κτηνοδών και απανθρώπων επιθέσεων που έστειλαν κύματα σοκ ε, σε όλη την Ευρώπη και ευρύτερα. Οι σκέψεις μας είναι με το γαλλικό λαό και ιδιαίτερα τις οικογένειες των θυμάτων. Αλλά η ανταπόκριση των Ευρωπαίων μέσω διαδηλώσεων και εκστρατιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έφερε πιο κοντά για να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου που αποτελεί και παραμένει πυλώνα της δημοκρατίας μας. Αξιότιμα μέλη. Η προτεραιότητά μας αρθρώνεται με βάση τρία κυρίως θέματα. Μία Ευρώπη ανταγωνιστική, ψηφιακή και αποφασιστική. Αυτά είναι θέματα που παίζουν μεγάλο ρόλο για τους απλούς Ευρωπαίους. Η Επιτροπή σας ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον κοινό πολίτη με δύο τρόπους. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει νομιμοποίηση, δηλαδή πρέπει να υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ ε, της Ένωσης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών. Το δεύτερο σκέλος των θεμάτων αφορά την πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το θέμα της νομιμοποίησης, θα ήθελα να σας μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και την διαφάνεια θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι ένα ιδιαίτερα πολύτιμο μέσο. Όχι μόνο μας δίνει ένα μοναδικό και πραγματικά ευρωπαϊκό κοινό χώρο για διαμεθοριακή συνεργασία, αλλά χορηγεί στους πολίτες τη δυνατότητα να επηρεάσουν ε, το θεματολόγιο της Ένωσης. Αυτή είναι μια σχετικά νέα διαδικασία και αντιμετωπίζουμε κάποιες προκλήσεις. Οπότε προσβλέπουμε στην έκθεση εφαρμογής της πρωτοβουλίας από την Επιτροπή τον Απρίλιο. Έχουμε πλήρη συνέστηση της σημασίας της διασφάλισης της διαφάνειας η οποία πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα με περισσότερη δυνατότητα για τους πολίτες να συμμετάσχουν ούτω ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης προς την Ένωση. Αυτό θα κατοχυρώσει την διαφάνεια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και θα ενισχύσει την νομιμοποίηση της Ένωσης. Να στραφώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε, το δικαστήριο πρόσφατα κατέληξε ότι το σχέδιο συμφωνία για την ένταξη, για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι σύμβατο με τις συνθήκες. Οπότε και τα τρία θεσμικά όργανα είναι σε δύσκολη θέση. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την Προεδρία μας για να διευκολύνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο και να συμφωνήσουμε για το πώς θα προωθήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα που θα επιτύχουμε. Όχι για τα ε, θεσμικά παζαρέματα στα παρασκήνια. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την, την Προεδρία μας για να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να βελτιώσουμε τη διοργανική συνεργασία με βάση τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που επέτυχε η Ιταλική Προεδρία θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσει θα λαμβάνονται στο πιο κατάλληλο επίπεδο. Γι' αυτό η Ένωση πρέπει να σεβαστεί τις αρχές της εκχώρησης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Και τα εθνικά κοινοβούλια ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά και πιστεύουμε βαθιά ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω στενής εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαι πεπισμένη ότι η στενή συνεργασία και η δημιουργία μια ευρεία συνένεση αναγκαία για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εφαρμόσουμε τη στρατηγική, το στρατηγικό θεματολόγιο για την Ένωση σε περίοδο αλλαγή. Από αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε ευγνώμονε και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή του και την ε, βούλησή του να διευκολύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να επιτύχουμε ομαλή πρόοδο για τα θέματα που μα ενδιαφέρουν από κοινού. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την Προεδρία μας για να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα για τον νομοθετικό προγραμματισμό για να έχουμε πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Με βάση τα ψήφια του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση τη διοργανικής συνεργασίας ελπίζουμε ότι θα στηρίξετε αυτή μας την πρωτοβουλία. Ο πρώτος ε, αντιπρόεδρος Τίμερμανς έχει εκφράσει την πρόθεσή του να υποβάλει πρόταση για την ε, μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση τη διοργανική συνεργασία για καλύτερη νομοθεσία του 2003 και προσβλέπουμε στη λήψη αυτή τη πρόταση Να αναφερθώ σύντομα και στο κράτο δικαίου. Λόγω τη σημασία που αποδίδει η Ένωση στο κράτο δικαίου στις, ε, διεθνεί διεθνείς τη σχέσεις είναι απόλυτα αναγκαίο να εφαρμόζουμε και στο εσωτερικό της Ένωσης πλήρως. Είναι θέμα προστασίας θεμελιώδους ευρωπαϊκής Αξία. Έχω συνέστηση ότι δεν έθιξα όλα τα θέματα. Αλλά προσβλέπω στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας και από αυτών στα οποία αναφέρθηκα ή και ευρύτερα φυσικά. Και τέλος θέλω να πω ότι προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας για το επόμενο εξάμεινο αλλά και, και περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο Γιώργ ε, Σέπφλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε εγώ προσωπικά και το ΕΛΚ. Νομίζω ότι σκεγγραφίσατε μια ευρεία εικόνα με όλα τα θέματα που κατά την άποψή σας είναι σημαντικά. Μετά την εμπειρία της Ουγγρικής Προεδρίας θα σας πω έχω να σας πω ότι τα γεγονότα πάντα θα σας εκπλήξουν. Θα σας εκπλήσουν, εκπλήσουν κάθε προεδρία, απρόβλεπτα γεγονότα. Είσαστε προετοιμασμένοι για τα απρόβλεπτα αυτά γεγονότα, διερωτώ με. Μετά τις επιθέσεις του Ιανουαρίου, προκύπτει ένα θέμα. Ήταν μία από τις από τις πιο απρόβλεπτες ε, προκλήσεις, ένα σοκ ε, που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίθεται το εξή ε, ερώτημα. ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Εσείς μιλήσατε για τη διαφάνεια. Νομίζω ότι υπάρχει μία πρόθεση από τη μία να έχουμε ασφάλεια και από την άλλη να έχουμε διαφάνεια. Τι προσέγγιση μπορούμε να έχουμε, τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε και ασφάλεια αλλά και διαφάνεια. Θέλω να σας πω, θέλω να ακούσω μεγάλο ενδιαφέρον την άποψή σας. Μπορείτε να κατολογήσετε για θέματα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και για την Ρωσία θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα έχετε τη ρωσόφωνη κοινότητα στην Λετωνία. Αν θέλετε να μιλήσετε και γι' αυτό, μπορεί να έχει σημασία. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε τι ποσοστό ρωσόφωνων έχουν την ηθαγένεια. Επίσης, είπατε ότι η πρωτοβουλία των πολιτών είναι χρήσιμο εργαλείο. Ως εισηγητής ενδιαφέρουμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Τι άποψη έχετε για αυτό το θέμα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει ένας τελικός μετασχηματισμός του ECI για να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο ε, επινοήθηκε τότε, την ε, εποχή της σύμβασης, της συνέλευσης. Είναι δύσκολο το θέμα και νομικός πώς υπάρχουν και τομείς που μπορεί να βελτιωθεί αυτή η πρωτοβουλία. Για τη μετανάστευση, τι άποψη έχετε. Είναι οξύ το πρόβλημα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο εσωτερικό δεν θα πρέπει να το πούμε μετανάστευση, αλλά έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζόμενων. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί λετονοί πολίτες ε, στα Βρετανικά νησιά. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν αρέσκονται να βλέπουν αυτούς τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω πόσο ψηλά είναι στους στόχους τους, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Επίσης υπάρχει και μετανάστευση από την Ουκρανία στη Λετωνία. Το θέμα είναι περίπλοκο. Τέλος. είπατε, μιλήσατε για τη σημασία του κράτους δικαίου, εδώ εντός το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστό. Ακούσαμε από τον Ιταλό Υπουργό, τον Σάντρο Γκότζι, για αυτή την ετήσια συζήτηση αυτών των γεγονότων στο Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι θα είσαστε προετοιμασμένοι για αυτή την ετήσια συζήτηση. Πώς σκοπεύετε να την οργανώσετε, ας πούμε, να την προωθήσετε. κυρία Μπρέσκο και μετά οι υπόλοιποι. Και μετά θα απαντήσει ο Υπουργός. Αν θέλετε να βάλετε ακουστικά, δεν νομίζω ότι, ότι καταλαβαίνετε Ιταλικά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και καλή δουλειά εσείς προσωπικά και η κυβέρνησή σας εν το συνόλο της. Αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια σημαντική χρονική στιγμή, γιατί τώρα ξεκινάει η νομοθετική δουλειά του Κοινοβουλίου, του νέου Κοινοβουλίου δηλαδή, και βεβαίως σημαντική γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή λόγω των επιθέσεων αυτών που έγιναν όχι μόνο φυσικός πώς, επιθέσεις προς Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και πολιτικές επιθέσεις. Μιλάμε για μια απειλή που επικρέμαται πάνω από την Ευρώπη. Να σας ρωτήσω, δεν πιστεύετε κι εσείς ότι η κυβέρνησή σας μετά από τα όσα έκανε η Ιταλική Προεδρία ε, θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας μέσα στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης, πιο ενισχυμένης συνεργασίας και ενδεχομένως να υπάρξει και μια θεσμική α, πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, προς την ευρωπαϊκή δηλαδή άμυνα και ασφάλεια. Ως σοσιαλίστρια και ως σοσιαλιστική ομάδα πιστεύουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Υπάρχει και μία γνωμοδότηση που την ετοιμάζουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία καταρχήν, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να την ξαναδούμε, να την αναθεωρήσουμε. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές, ούτω ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο για τους πολίτες να τη χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, εάν έχετε κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί λιγάκι αυτή η πρωτοβουλία ούτω ώστε να δώσουμε απάντηση σε πολλούς πολίτες που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά δυσκολεύονται γιατί έχει πολλές πρακτικές δυσκολίες αυτό το εργαλείο. Είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουμε υπογραφές, ούτω ώστε να παρουσιαστούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Τρίτον, το θίξατε και αυτό. Αλλά θέλω να μου πείτε πώς σκοπεύει η Προεδρία να κινηθεί, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή, αλλά και το Συμβούλιο αυτό καθεαυτό, για αυτό το θέμα, το οποίο είναι το εξής. Είναι εγγεγραμμένο αυτό το σημείο στην ε, συνθήκη, αλλά για το οποίο έχουν γίνει παρατηρήσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πολλές παρατηρήσεις, σημαντικότατες. Τι είδους πρωτοβολία θα πρέπει να πάρετε μαζί με άλλα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε να υπάρξει μια πρόοδος στην επικύρωση της σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε λίγο θα έρθει εδώ ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μεταξύ άλλων θεμάτων θα μας μιλήσει για τη συμφωνία την διαθεσμική. Θα μπορούσατε κι εσείς να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για την κατεύθυνση που σκοπεύετε να ακολουθήσετε για αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω κύριε Υπουργέ. για τη σύντομη παρουσίασή σας. Και τον Πρωθυπουργό σας για την ομιλία του στο Στρασβούργο, που ήταν και λακωνική, αλλά και πολύ σημαντική με πολύ έντονη έτσι, ευρωπαϊκή χρειά. Λόγω της ε, γεωγραφικής θέσης της Λετωνίας και της δραματικής ιστορίας και του γεγονότος ότι μπορεί να συμμετάσχει τώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ας πούμε, θα ήθελα να σας θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Για την πρωτοβουλία των πολιτών μας, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Η κρίση που μαστίζει αυτό το εργαλείο δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Ε, συχνά παραπονιόμαστε για τη χαμηλή προσέλευση σε ευρωπαϊκές εκλογές και προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να βελτιώσουμε αυτό το πρόβλημα. Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Η εκστρατεία One of Us, ένας από εμάς, είχε υποστήριξη από 1,7 εκατομμύρια πολίτες από διαφορετικές χώρες. Η κρίση συνίσταται στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πολύ δογματική προσέγγιση απέναντι σε αυτό το εργαλείο. Ο Επίτροπος Τίμερμανς έχει μια πολύ νομικήστική προσέγγιση. Δεν, το, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι πολίτες αδιαφορούν για αυτή την πρωτοβουλία. Αντίθετα, ενδιαφέρονται, την υποστηρίζουν. Και τη χρησιμοποιούν κιόλα. Ευρέω. Αλλά μπλοκάρεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν συνεχεία, η πρωτοβουλία αυτή. Εξού και λοιπόν και το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι η προσέγγιση της Λετωνικής Προεδρίας για το θέμα αυτό, τι μπορούμε να περιμένουμε από εσά Μπορείτε να μας βοηθήσετε για να απεμπλακεί το πρόβλημα που μπλοκάζει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, λοιπόν, τελευταίος ο Χάουρεγγι. Δεν υπάρχει άλλος να θέλει το λόγο. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Έχω δύο ερωτήματα να σας θέσω σχετικά με την Επιτροπή μας. Πρώτον, και κυρία Μπρέσο και εσείς αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Ε, σε ό,τι αφορά την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν. Θα σας θυμίσω κάποιες ημερομηνίε. Πρόκειται για απόφαση που προέρχεται από τη Συμφωνία της Λισαβόνας, που ετέθησε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2009. Το καλοκαίρι του 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το πλαίσιο αυτής της ένταξης. Για τέσσερα χρόνια η Κομισιόν και το Συμβούλιο διαπραγματεύθηκαν με το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου τους όρους με τους οποίους θα γινόταν η ένταξη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν ε, είπε ότι το πλαίσιο που διαπραγμάτευσης ε, είναι ασύμβατο. Είναι συμβατό υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν πέντε τροποποίησεις σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή η διαπραγμάτευση να ξαναρχίσει. Διότι αν ε, ε, σεβαστούμε αυτές τις πέντε παρατηρήσεις του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να γίνει η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε προβλεπόταν συνθήκη της Λισαβόνας ε, και γι' αυτό το λόγο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί. Θα πρέπει να δούμε αν η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάδει με, την, με το, τη συμφωνία. Για παράδειγμα, το στρατιωτικό μας προσωπικό όταν δράσει οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή σε ένα μέρος του κόσμου. Πρέπει να μην μείνει στο σιρτάρι αυτό το θέμα. Δεύτερον, ε, χάρη στην ε, ε, συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει ερευνητικές επιτροπές. Ο κανονισμός όμως του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε το 2012 και που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των επιτροπών ε, έχει ε, μπλοκαριστεί γιατί η Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, εξέφρασαν επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία της έκθεσης του Κοινοβουλίου. Ήδη εμείς εδώ έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε το θέμα αυτό προκειμένου να ζητήσουμε από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο να ξαναξεκινήσει ο τριμερής διάλογος για αυτό το ζήτημα. Αυτή τη βδομάδα θα συναντηθώ με μια εκπρόσωπο της κυβέρνησής σας ακριβώς για να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Και θα ήταν σημαντικό και εσείς να έχετε υπόψη ότι η Λετωνική Προεδρία θα μπορούσε πραγματικά να οθήσει, να προωθήσει αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ζητήσω τώρα ε, από την κυρία Υπουργό να απαντήσει. Το πήρες. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Σόπλιν. Σε αυτή τη αφορά τα απρόσμενα γεγονότα και απρόλεπτες καταστάσεις για τις οποίες θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ε, σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και διαφάνειας. Η... Πάντοτε λέμε ότι είμαστε, έχουμε πει μάλλον επανειλημμένως ότι ε, ε, είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδου γεγονότα. Σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και διαφάνειας, οι στρατηγικέ κατευθύνσεις γραμμές που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 και 27 Ιουνίου ε, πέρσι ε, θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την εσωτερική στρατηγική ασφάλειας ε, μέχρι το μέσο του 2015. Αυτό προβλεπόταν. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια λοιπόν της Λετωνικής Προεδρίας και για μας θα είναι προτεραιότητα. Τα πρόσφατα γεγονότα στο Παρίσι απέδειξαν πόσο σημαντική είναι αυτή η εργασία. Η Λετωνική Προεδρία αναμένει την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Έχει ε, ανακοινωθεί ότι θα είναι έτοιμη την Άνοιξη, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Η αναθεώρηση της εσωτερικής στρατηγικής ασφάλειας θα βασιστεί σε αυτή την ανακοίνωση. Πρόσφατα υιοθετήσαμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, ανανέωση της στρατηγικής αυτής. Η... Τα βασικά στοιχεία αυτής της αναθεωρημένης στρατηγικής ε, θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός και ορισμός των ε, απειλών, ε, η συνεπής και διαστομένη προσέγγιση, η σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η εφαρμογή. Για να εξασφαλίσουμε την πιο διευρυμένη δυνατή στήριξη αυτής της προσέγγισης. Η Προεδρία αναμένει και ελπίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει θετικά. Σε ό,τι αφορά την μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στρασβούργο το θέμα των, της μετανάστευσης. Το Συμβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για την συνεχιζόμενη μαζική άφηξη μεταναστών στη Μεσόγειο. το μεταναστευτικό βάρος ε, αυξάνεται και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν είναι τόσο πολλοί οι Ουκρανοί που έρχονται στη Λετωνία. Παρ' όλα αυτά ε, έχουμε δει συχνά ε, λάθρομετανάστευση και μέσω ε, πλοίων φαντασμάτων. Θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, απτά μέτρα και να υπενθυμίσουμε ότι η Task Force της Μεσογείου ε, ε, ε, είχε προωθήσει την ενίσχυση των συνόρων ε, και τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της ε, λαθρομετανάστευσης ως προτεραιότητες. Οπότε ε, αυτές οι προτεραιότητες ήδη ε, ε, ε αυτές ήδη υλοποιούνται και ο, η, η, εφαρμογή του τρίτονος ε, της επιχείρησης τρίτων ε, το δείχνει αυτό. Για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δεν έχουν ασχοληθεί τίποτα περισσότερο. Είναι η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να διατηρηθεί. κ. Σουεπφλίν και η κυρία Μπρέσο και ο κύριος Γιάντοφσκι μίλησαν για την Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία των Πολιτών. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, αλλά και το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες των Πολιτών είναι σημαντικό βήμα προκειμένου να εμπλακούν οι πολίτες στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο αναμένει με ανυπομονησία την έκθεση της ε, Κομισιόν για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Θα είναι έτοιμη τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια λοιπόν της Λετωνικής Προεδρίας. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συζητήσει όλες τις νόμους που υπάρχουν για την βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος της ε, πρωτοβουλίας. Ε, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη και, την, ε, και του Κοινοβουλίου και την ε, γνώμη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Το Συμβούλιο θα εξετάσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, όλες τις ε, προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος, για παράδειγμα για την αύξηση της γνώσης πλευράς των πολιτών, της ύπαρξης αυτής της δυνατότητας, ε, Καθώ επίση και τη διευκόλυνση σε ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Είναι πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών για την βελτίωση τη ε, δημοκρατία και της συμμετοχή δημοκρατία πιο συγκεκριμένα. Να σας πω ποιε είναι οι δικέ μα εμπειρίε πριν από μερικά χρόνια στη Λετωνία δώσαμε τη δυνατότητα στους πολίτες μας ε, να συλλέξουν 10.000 ηλεκτρονικές υπογραφές προκειμένου να ξεκινήσουν εθνική πρωτοβουλία πολιτών ε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κίνηση κοινωνίας μας. Όταν συλλεχθούν 10.000 ε, υπογραφές, ηλεκτρονικές υπογραφές για ένα οποιοδήποτε θέμα, το Εθνικό μας Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να συζητήσει το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι πολύ σημαντικό και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε αυτή η έκθεση σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το σύστημα. και να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που παρέχει. Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, η Προεδρία καλωσορίζει την απόφαση εκείνης διαλόγου για το θέμα αυτό στο, στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Ερώτηση κυρία Μπρέσο και του κυρίου Χαουρεγκή. Ε, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την σύμβαση ε, προβλέπεται από την συνθήκη της Λισαβόνας και αποτελεί κλειδί για την ολοκληρωμένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσεκτικά εξετάζουμε την γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει ότι το προσχέδιο συμφωνίας ε, δεν είναι συμβατό με τις συνθήκες. Το δικαστήριο έχει εντοπίσει συγκεκριμένα αρκετά σημεία ε, ασυμβατότητας. Ε, η κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλεια είναι ένα από αυτά. Η γνωμοδότηση βέβαια του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζει ούτε ακυρώνει ε, το, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6.2 του, της Συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει έναν ε, ε, επικοδομητικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία προετοιμάζει την ε, πρώτη επίσημη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πρέσβεων για το πώς θα προχωρήσουμε. Θα αποτελέσει μία από τι προτεραιότητε μας λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων από το πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του, της, του εποπτικού έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρόβλημα είναι ότι οι εξελίξεις τώρα έχουν ε, ε, δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα οποία δεν έχουμε λύσει ακόμα, όπως για παράδειγμα πρόσβαση σε ε, έγγραφα, θέματα κυρώσεων για, την, μη, για το μη σεβασμό των πορισμάτων, το Συμβούλιο από την άλλη μεριά ε, είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο αν υπάρχουν καινούριε προτάσεις. Σε ό,τι φορά την Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής δεν θα ήθελα να επισέλθω σε, στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ύπατης εκπροσώπου. Ε, εμείς από τη μεριά μας θα συνεργαστούμε στενά με την ύπατη εκπρόσωπο για όλα αυτά τα θέματα μεταξύ αυτών Ρωσία και Ουκρανία. Όπως επίσης και στη σχέση μας με την νότια διάσταση. Χτες ε, έλαβε χώρα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και συζητήθηκε το θέμα της Ρωσίας. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αλλάξει. Το σημαντικό είναι το, το Συμβούλιο να εκφράζεται με μια φωνή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι βασικές ερωτήσεις σας. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ήλπιζα να το θίξουν οι συνάδελφοι. Κατά την Ιταλική Προεδρία υπήρξε αυτή η ομάδα εργασίας φίλη της Προεδρίας επιθεσμικών θεμάτων πώς η Ευρώπη δηλαδή θα γίνει πιο αποτελεσματική και για μια προσεχή διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία. Αναφέρθηκε η πρόθεση το Δεκέμβριο να υπάρξει μια διακήρυξη, να δεσμευθούν όλα τα θεσμικά όργανα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τελικά δεν υπεγράφει. και ίσως και το Κοινοβούλιο γι' αυτό. Ερώτηση λοιπόν. Κατά την Προεδρία σας θεωρείτε ότι θα τα καταφέρουμε τα τρία θεσμικά όργανα να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε μία αναθεώρηση και βελτίωση της διοργανικής συμφωνίας του 2003 για καλύτερη νομοθεσία. Έχετε τέτοια σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Υπουργός. Το συζητήσατε σήμερα έτσι δεν είναι και με την Ιταλική Προεδρία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία που επετέλεσε η Ιταλική Προεδρία. Και για το μέλλον τώρα. Βεβαίως προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Επιτροπή σας για θέματα ενωσιακού συμφέροντος. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Ταλικής Προεδρίας για διοργανικό προγραμματισμό για να διευκολύνουμε τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Ένωσης σεβόμενοι βεβαίως ε, το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Και το Συμβούλιο δεσμεύεται να ενισχύσει τη διοργανική συνεργασία διασφαλίζοντας πιο αποτελεσματική διαδικασία και καλύτερη νομοθεσία. Η διοργανική συμφωνία του 2003 Ακριβώς στα πλαίσια των τριών προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτά τα θεσμικά θέματα για να ενθαρρύνουμε, ή συγγνώμη, για να βασιστούμε στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της Ιταλικής Προεδρίας. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόταση για να διαπραγμάτευσε τη συμφωνία του 3 για καλύτερη νομοθεσία και αυτό αντιμετωπίστηκε με ευρεία συνένεση από τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή λοιπόν θα υποβάλει την πρότασή της και μετά η Προεδρία μας θα κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά για την αναθεώρηση αυτής της διοργανικής συμφωνίας του 2003 από πλευράς του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, είχαμε την πρόθεση ως ΑΦΚΟ να επισκεφθούμε τη Ρήγα και το συζητήσαμε ε, και τελικά καταλήξαμε 18 με 20 Μαρτίου. Πρόθεσή μας βεβαίως είναι να έρθουμε σε επαφή με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης αλλά και ευρύτερα με εκπροσώπους της κοινωνίας, το κοινοβούλιο και ίσως και μερικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ή και με άλλους φορείς που εσείς θα θεωρούσατε ότι είναι σημαντικό να δούμε. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή και θα μας βοηθήσετε έτσι δεν είναι για να οργανώσουμε αυτή την επίσκεψη. για να μπορέσουμε να δούμε και τι επιτυχίες έχουν σημειώσει οι Λετονοί τις τελευταίες δεκαετίες για ένα καλύτερο μέλλον, για σταθερότητα και πώς έχουν ωφεληθεί από την ένταξή τους στην Ένωση. Θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που είναι τμήμα αρμοδιοτήτων μας. Και θα βασιστούμε πολύ στην εργασία σας. Πρόεδρος, βεβαίως, μα με μεγάλη χαρά θα σας καλωσορίσουμε στη Ρήγα. και θα σας βοηθήσουμε, ούτω ώστε να είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψή σας, ε, είναι πολύ σημαντικό να συναντηθείτε όχι μόνο με εκπροσώπους της κυβέρνησής μας, με κοινοβουλευτικούς, εκπροσώπους μη όμικρον κοινωνικών εταίρων, ως ε, πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μας είμαι πεπισμένη ότι και το Κοινοβούλιο θα σας υποδεχθεί, θα έχετε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ότι θα γίνετε δεκτή και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και μου είπαν ότι και εκείνοι ε, θέλουν πολύ να σας δουν. Νομίζω πως θα είναι μια πολύ καλή συνέχιση των σημερινών μας συζητήσεων και βεβαίως πρόθεσή μας το προσεχές εξάμεινο είναι να συνεργαστούμε πολύ στενά με την Επιτροπή σας. Θέλουμε στενότερους δεσμούς με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό τμήμα αυτό της Προεδρίας μας, των δεσμεύσεών μας. Και η ανταλλαγή απόψεων καταδεικνύει ότι συμμεριζόμεθα πολλές προτεραιότητες και όραμα για τη θεσμική συνεργασία, για τη διαφάνεια και πολλά άλλα. Πολύ σημαντικά. Προσβλέπουμε λοιπόν στη στενή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αλλά και μετά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Συνάδελφοι, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ε, μισή ώρα και πάνω που έχουμε για να προτάξουμε το 13 για να συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Ραμόν Χάουρεγγι. Ενημερώσαμε τους σκιώδεις και πάνω από τους μισούς ε, τους βλέπω εδώ, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην συζήτηση. Ξέρετε ότι είναι ειδική περίπτωση έκθεσης που συζητήσαμε στην προηγούμενη θητεία και είχαν γίνει και οι τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό αλλά δεν καταλήξαμε δεν ολοκληρώσαμε κατά την προηγούμενη θητεία το προηγούμενο κοινοβούλιο είχε ψηφίσει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια κατά την τρέχουσα λοιπόν θητεία θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα για να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσει, όχι να αρχίσουμε από το μηδέν και ζητήσαμε και από, το, από τη διάσκεψη των Προέδρων να ε, λάβει απόφαση ότι είναι δυνατόν να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, να συνεχιστούν. Και να δώσω το λόγο στον Ραμόν Χάουρεγγι, που είναι ο νέος εισηγητής που αντικατέστησε τον Ντέιβιτ Μάρτιν, ο οποίος δεν είναι πλέον μέλος της Επιτροπής μας. Παρακαλώ κύριε Χάουρεγγι. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, η υπόθεση αυτή έχει αρκετό παρελθόν στο Κοινοβούλιο. Να σας ενημερώσω λοιπόν για να συζητήσουμε κάπως πιο εμπεριστατωμένα το θέμα. Η δυνατότητα δημιουργίας εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει δυνατότητα να φέρει σε πέρας μία από τις πιο χαρακτηριστικές λειτουργίες ενός πραγματικού κοινοβουλίου, η δημιουργία εξεταστικών των πραγμάτων επιτροπών. Και ε, ξεκίνησε αυτή η δυνατότητα ε, από την ε, συνθήκη του Μαστρίχτ το 1993. Αυτή ήταν η πρώτη δυνατότητα. Δεν ήταν κανονισμός λοιπόν. Ήταν απλώς μια διοργανική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής για να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το δικαίωμα δημιουργίας εξεταστικών επιτροπών έπρεπε να υλοποιείται. Αυτό συμφωνήθηκε το 1995, αυτή η διοργανική συμφωνία λοιπόν. Αυτή η συμφωνία ακόμη διέπει τη δημιουργία εξεταστικών επιτροπών, εξακολουθεί να ισχύει. Κατά την διάρκεια λοιπόν λειτουργίας αυτής της συμφωνίας, σχεδόν 20 χρόνια, στο Κοινοβούλιο υπήρξαν τρεις εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές για τρία πολύ διαφορετικά θέματα. Πρώτη, απάτες ε, του ΦΠΑ και απάτες για τον, ΦΠΑ και τους τελειωνιακούς δασμούς το 97 για την περίφημη υπόθεση των τρελών αγελάδων επίσης το 97 και για την ε, κατάρρευση μιας ε, ασφαλιστικής εταιρείας το 2007. Όμως, η συνθήκη του Λισαβόνας, επιχειρώντας επανεξισορρόπηση εξουσιών μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, χορηγώντας περισσότερη εξουσία στο Κοινοβούλιο, ενίσχυσε την πολιτική σημασία του Κοινοβουλίου και του χορήγησε πολύ συγκεκριμένη εντολή για τη δημιουργία μέσω δικαιώματος πρωτοβουλίες που δεν έχουμε για κανένα άλλο θέμα. Χορήγησε λοιπόν στο Κοινοβούλιο η συνθήκη της Λισαβόνας τη δυνατότητα να δημιουργήσει κανονισμό για να ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας αυτών των επιτροπών. Και λοιπόν το Κοινοβούλιο με εισηγητή τον David Μάρτιν το 2010 λοιπόν ο οποίο όμως τώρα είναι συντονιστή στην Ίντα και άρα δεν είναι εδώ στην ΑΦΚΟ. Το Κοινοβούλιο λοιπόν εξεπώνησε την πρώτη έκθεση έναν κανονισμό που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2012 και δημιούργησε μια πολύ πιο αναλυτική νομοθεσία, λεπτομεριακή θα έλεγα, για τις δυνατότητες, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δημιουργεί επιτροπές έρευνας. και για να έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει ενεργά με πολύ πιο ευρύ τρόπο μέσω της διοργανικής συμφωνίας. Η έγκριση λοιπόν το Μάιο του 2012 αυτού του κανονισμού όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος προκάλεσε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα τα οποία προέβαλαν ε, αρκετές και νομικές και πολιτικές αντιρρήσεις για τις εξουσίες που ήθελε να ε, αναλάβει το Κοινοβούλιο μέσω αυτών των εξεταστικών επιτροπών. Τώρα για να μην πω πολλά. Οι αντιρρήσεις αυτές, νομικές και πολιτικές, για τα, αυτά που πρέβλεπε το 5, το 8, το 12 και το 14. Συγκεκριμένα. Τις εξουσίες που χορηγούσε στον εαυτό το κοινοβούλιο να διερευνήσει, παρά το ότι θα μπορούσε να υπάρχει δικαστική έρευνα, κάτι που απαγορεύει στην Λισαβόνα. Και εδώ έχουμε ένα πρώτο πρόβλημα. Διότι Εάν υπάρχει δικαστική έρευνα για ένα θέμα, τα άλλα δύο θεσμικά όργανα λένε δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να φτιάξει μια ε, εξεταστική επιτροπή. Άρα το θέμα είναι ποιο θα αποφασίσει. Εάν το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να έχει μια τέτοια επιτροπή που να διερευνά ένα θέμα. Διότι μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να διακόψει, να αναστείλει μια τέτοια διαδικασία. Δεν μπορεί να το αποφασίσει κάποιο δικαστήριο. Κανένα δικαστή, καμία χώρα είναι απόλυτο δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα θέμα επίσης εμπιστευτικότητα των εγγράφων που μπορεί να απαιτήσει από άτομα ή από κράτη το Κοινοβούλιο. Πώς λοιπόν θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα είτε ατομικά είτε ευρύτερα τα δικαιώματα στην ιδιωτική σφαίρα. Πώς δηλαδή θα διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των εγγράφων που πρέπει να είναι μυστικά. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι όντως θα είναι στην πράξη. Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα με το τι αρμοδιότητα έχει το Κοινοβούλιο όταν έρθουν κάποιοι πάλι εδώ ή όταν δεν έρθουν και έχουν κάποιο λόγο να μην έρθουν σε ποιο θα την εξηγήσουν δηλαδή έχει ένα πρόβλημα με τις εξουσίες που ανέθεσε στον εαυτό του το Κοινοβούλιο να μπορεί να πει ούρμπι ετόρβε σε οποιοδήποτε πολίτη και οποιοδήποτε φορέα ότι πρέπει να παρευρεθεί, να κλητευθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Και επίσης, τι κυρώσεις μπορούν να επιληθούν σε όσους δεν παρευρεθούν, δεν προσέλθουν. Διότι ε, με σωστή νομική αντιμετώπιση και το Συμβούλιο και η Κομισιόν, σωστή κατά τη γνώμη μου, Μα λένε ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσει. Και επιπλέον οι δυνατότητες κυρώσεων, ποινικών ή όχι, στι διάφορες χώρες είναι πολύ διαφορετικές. Και διαφορετικές επίσης ρυθμίσεις όσον αφορά το εάν και κατά πόσον υποχρεούνται κάποιοι να προσέλθουν ενώπιον μιας εθνικής ή ευρωπαϊκής εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Αυτά λοιπόν είναι ευαίσθητα θέματα. Γι' αυτό υπήρξε αδίέξοδο. Και αυτό όθησε το Κοινοβούλιο να αποφασίσει να εγκρίνει την αρχή του κανονισμού αλλά να αφήσει για την επόμενη θητεία, δηλαδή για την παρούσα θητεία που προέκυψε από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου το μέλλον αυτού του κανονισμού. Και καταλήγω. Καταλήγω. Εδώ βασίζονται λοιπόν οι προτάσεις που υποβάλλω στην Επιτροπή μας για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε την εξέταση του θέματο αυτού. Πρώτον, να θέσω ένα θέμα πολιτικό αρχής, που είναι πολύ σημαντικό να εμείνουμε επ' αυτού. Το Κοινοβούλιο έχει το δικό του κανονισμό τον οποίο να αποφάσισε με βάση τη δική του πρωτοβουλία, όπως καθορίζει η συνθήκη του Λισαβόνα, που του χορηγεί τη δυνατότητα να δημιουργεί τέτοιε επίτροπε όταν ε, προκύψει μία μη εφαρμογή ή μία κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων από ένα οργανισμό, ένα κράτος ή ακόμη, μπορώ να προσθέσω, και από ιδιώτες, από επιχειρήσεις για παράδειγμα δηλαδή εννοώ, που δεν εφαρμόζουν επαρκώς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχει λοιπόν δυνατότητα να δημιουργεί επιτροπές ερευνητικές, ad hoc. Είναι θέμα αρμοδιότητας ενός κοινοβουλίου. Αυτό έχει να κάνει με την κυριαρχία και την ε, πολιτική φύση. Αυτό λοιπόν διακυβεύεται. Δεν μπορεί το κοινοβούλιο να εγκαταλείψει αυτή την αρμοδιότητα. Να έχει λοιπόν την επαρκή ad hoc νομοθεσία για να εφαρμόσει αυτό το δικαίωμα που είναι απόλυτα φυσιολογικό και χαρακτηριστικό για οποιοδήποτε κοινοβούλιο μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατικό. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι οι αντιρρήσεις που λάβαμε από τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής μέσω επιστολής που απεστάλλει στο Γενικό Γραμματέα του σώματός μας πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι έχουν κάποιο νομικό και πολιτικό περιεχόμενο που πρέπει να εξετάσουμε. Κατά τη γνώμη μου, και θέλω να σα ενημερώσω για τη γνώμη μου, αυτό είναι πιο σημαντικό από το να έχουμε έναν κανονισμό, γιατί το πιο σημαντικό είναι η πολιτική και νομική συζήτηση θα καταλήξει σε κάποια συνένεση. Και αυτή είναι η βούλησή μου. Θα ήθελα οι σύντροφοί μου από τις άλλες πολιτικές ομάδες θα ήθελα να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει διάλογος για να καταλήξουμε σε ένα λογικό κανονισμό. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να μετριάσει τις απόψεις τους. Υπάρχουν κάποια νομοτεχνικά θέματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και για να καταλήξω, να καταλήξω στο τελικό μου συμπέρασμα. Ζήτησα από τη Λετωνική Προεδρία να συζητήσουμε με το θέμα αυτό εδώ και λίγα λεπτά όταν ε, συζητούσαμε με την Υπουργό, επίσης το συζητήσαμε και ε, υπενθυμίζω ότι είπα ότι σε δύο μέρες θα συναντηθώ με εκπροσώπους της... Συγγνώμη, σε τρεις μέρες, την Παρασκευή. Θα συναντηθώ με εκπροσώπους της Λετωνικής Προεδρίας για να ε, τους πείσω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουν και να συνεργαστούμε. Και ανάλογα με την απάντηση που θα μας δώσουν, ίσως να είναι αναγκαίο κυρία Πρόεδρε, εσείς να απαιτήσετε από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να επανέλθουμε σε έναν τριμερή διάλογο, πρώτα απ' όλα σε πολιτικό επίπεδο, για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και μετά να δούμε και αν θα μπορούσαμε να έχουμε τεχνικό διάλογο για να λύσουμε αυτό το θεμελιώδε θέμα του επόμενου μήνε. Γιατί είναι μια δημοκρατική εξουσία του Κοινοβουλίου μα και ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Βίλαντ. Από πλευρά ΣΕΛΚ. Ευχαριστώ. τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία του. Με πολύ σαφή τρόπο παρουσιάζει την προϊστορία του θέματος αυτού και τη συνοψίζει. Ο Νάρσος Μάρτιν ασχολήθηκε πολύ με το θέμα αυτό. Είχαμε επίσης ε, συζητήσεις ε, επανειλημμένα του εισηγητή και των σκιωδών με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και διαπιστώσαμε ότι το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα αδιάλακτο για το θέμα αυτό. Και εξεπλάγει. Πρέπει να το πω ανοιχτά. Εξεπλάγει γιατί και η Επιτροπή είναι αδιάλακτη. Το αντικείμενο μιας εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι πολιτικό. και να προκύπτουν και θέματα πολιτικών, προεκλογικών σκοπιμοτήτων, γιατί προτείνονται κάποια θέματα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοια. Το θέμα είναι πώς θα εργαστεί μια εξεταστική επιτροπή. Το θέμα της συνεργασίας των πολιτικών οργάνων είναι πάντα πολιτικό θέμα και προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτό το θέμα. εξεταστική επιτροπή, μια εξεταστική επιτροπή δεν πρέπει να είναι χάρτινος τίγρης. Έχω συμμετάσχει σε επιτροπές ε, έρευνας και διαπίστωσα ότι είναι πολύ περιορισμένες δυνατότητές μας. Και υποστηρίζω τον εισηγητή που λέει ότι πρέπει να δείξουμε ευελιξία. Αλλά υπήρξε ευρία απόφαση του Κοινοβουλίου για να υπάρχει ευελιξία. 95%. 95% είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευελιξία και καλή θέληση από πλευρά Κοινοβουλίου. Αλλά από πλευρά Επιτροπή και Συμβουλίου δεν είδαμε και πολύ καλή θέληση και ευελιξία. Πρέπει στο μέλλον να δείξουν περισσότερη καλή θέληση. Στην έκθεσή μα που εγκρίθηκε λοιπόν όπως είπαμε ευρεία πλειοψηφία, περιέχονται και μερικέ κόκκινε γραμμέ. Και πρέπει να παραμείνουν κόκκινε γραμμέ. Και τι σημαίνει αυτό, ποιε είναι αυτέ. Πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε όλα τα έγγραφα. Και βεβαίως, βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε ευρύτερα, ε, πέρα από, την επιτρο... από τις ε, οδηγίες διαφάνειας. Δηλαδή το κοινοβούλιο μπορεί να βλέπει έγγραφα, το οποίο δεν θα πρέπει να δει το ευρύ κοινό ή κάποιος λομπίστας. Πρέπει να μπορεί να δει πολύ περισσότερα έγγραφα. Και αυτό δεν καταλαβαίνω την επιφυλακτικότητα. Για μένα είναι αναμφίβολο ότι όσοι εμφανίζονται, όσοι προσέρχονται ενώπιον εξεταστικών τροπών πρέπει να πει την αλήθεια. μπορούμε να παρακαλέσουμε την ε, υπηρεσία έρευνά μα να μα πει σε ποια κράτη-μέλη υπάρχουν τέτοιε επιτροπέ, σε ποια κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κλητεύσει και σε ποια κράτη-μέλη. Οι καταθέσεις τους ενώπιον εξεταστικών επιτροπών γίνονται ε, χωρίς ε, να χρειαστεί, ε, όχι με όρκο, αλλά παρόλα αυτά, αν αποδεχθούν ψευδείς, υπάρχουν δυνατότητες κυρώσεων. Και σε ποια κράτη-μέλη υπάρχουν δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα η Επιτροπή να υποβάλει σε όρκο τους εμφανιζόμενους, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν αντίστοιχες κυρώσεις. να μας πούνε τι δυνατότητες έχουμε. Να μάθουμε εάν υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά εφόσον σε κάποιες χώρες υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων, τότε θα πρέπει να υπάρχουν ε, τουλάχιστον ισοδύναμες δυνατότητες κυρώσεων ή τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα απειλής τέτοιων κυρώσεων για οποιονδήποτε καταθέσει ψευδός ενώπιον ε, Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Και θα ήταν σκόπιμο πιστεύω να πούμε σαν κράτος μέλος εάν εσύ ο κράτος μέλος δεν θέλεις να στείλεις ένα υπάλληλό σου τότε τουλάχιστον πρέπει να το αιτιολογήσει. Και η αιτιολόγηση βεβαίως ε, δεν, μπορεί, δεν είναι αναγκαίο να είναι γραπτή αυτή η εξήγηση. Μπορεί να έρθει ένα υπουργό και να μα πει γιατί δεν πρέπει να έρθει ένα υπάλληλο. σω γιατί το απαγόρευσε. Ο επίτροπος Σεύκοβιτ, που ήταν αρμόδιος στι προηγούμενες ε, συζητήσεις που κάναμε δεν ήθελε να κάνει αυτή τη διάκριση διότι οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή επιτροπή βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν εδώ και είναι πολύ πιο κοντά σε εμά από ότι πάλι από τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό είναι λογικό να υπάρχει υποχρέωση ιδεολόγησης πολύ ψηλότερη για έναν ε, υπάλληλο τη Κομισιόν, πολιτικά και νομικά, από ό,τι αιτιολόγηση για το γιατί δεν προσέρχεται ένας εθνικός υπάλληλο. Ποτέ δεν κατάλαβα. Γιατί η Κομισιόν εκνευρίστηκε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να κάνει αυτή τη διάκριση. Και θα πρότεινα να διατηρήσουμε αυτή τη διάκριση. Ναι, ευελιξία στο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε κόκκινες γραμμές, δηλαδή σε σημεία στα οποία είμαστε ανυποχώρητοι μεταξύ εισηγητή και σκιωδών. Δεν χρειάζεται να τα ανακοινώσουμε όλα αυτά βεβαίως δημόσια, ποιες θα είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Μπορείτε να είστε σίγουροι κύριε εισηγητή ότι για ορισμένα θέματα θα βαλέψουμε περισσότερο, για άλλα λιγότερο, αλλά να είστε σίγουρος κύριε εισηγητά ότι αν κάποιε κόκκινε γραμμέ δεν περιέχονται, τότε μπορούμε να πούμε καλύτερα να μην υπάρξει συμφωνία. Και καλύτερα τότε να πούμε δεν υπήρξε συμφωνία και να καταδείξουμε του υπεύθυνου και να καταλήξουμε και να δηλώσουμε ότι δεν υπήρξε καλή διάθεση από πλευρά όλων, αλλά δεν ήταν δυνατόν να καταλήξουμε συμφωνία. Μάιτε Ρουίθ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πολύ σαφή παρουσίαση. Ας είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να καταφέρουμε να διαθέτουμε αυτό το εργαλείο και να μην χάσουμε τη δυνατότητα θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε με εντιμότητα έτσι ώστε να βρούμε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή που θα ε, δώσει σάρκα και οστά σε αυτό το εργαλείο. Ο κ. Χαουρική έχει δίκιο που λέει ούτε ότι δεν μπορούμε να απαρνηθούμε αυτό το όργανο ρεαλιστές. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ή όλα ή τίποτα. Ας, ε, θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή ε, γιατί πρόκειται για ένα εργαλείο που χρειαζόμαστε όπως και άλλα εργαλεία τα οποία χρειάζεται το Κοινοβούλιο προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο του της ε, παρακολούθησης και του εντοπισμού των κακών πρακτικών σε διάφορα θεσμικά όργανα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή, θα συνεργαστούμε και θα τον βοηθήσουμε ε, σε ό,τι χρειαστεί για να καλυφθεί το νομικό κενό. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ο Μαξ Άντερσον είναι εδώ. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πράσινοι διάβασαν το έγγραφο. Μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και υποστηρίζουμε τον εισηγητή. Συνεχίστε έτσι και θα είμαστε με το μέρος σας. Οι επόμενοι δύο μιλητέ δεν είναι εδώ και ο Σόλτς δεν είναι. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Πριν από δύο λεφτά η καρέκλα σας ήταν άδεια, αλλά να σας. Ήρθατε. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό αυτό το δικαίωμα του Κοινοβουλίου, το δικαίωμα να συστήσει εξεταστικές επιτροπές. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη Διαθεσμική Συμφωνία. Δεν ήμουν από την αρχή της συζήτησης. Εξήγησε ήδη ο εισηγητής κατά πόσο πιστεύει ότι θα συμφωνήσει το Συμβούλιο για να συστήσουμε τέτοιες εκταστικές των πραγμάτων επιτροπές. Ο κύριος Βίλαν ανέφερε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα των κρατών μελών καθώς και της Επιτροπής. Έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι μπορεί να κάνουν αυτές οι εκταστικές επιτροπές. αν δεν εξετάζουν μόνο το έργο της ε, Κομισιόν αλλά και το έργο των κρατών μελών. Ίσως θα πρέπει να μπούμε εδώ σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας στο μέλλον, ούτως ώστε να μπουν και περισσότερες ε, λεπτομέρειες στην έκθεση αυτή που συντάξατε. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Αν όχι, η πρόταση του Ραμόν Χαουρέγγι είναι ότι θα γίνει την, Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή η συνάντηση, έτσι. Αυτή την Παρασκευή θα γίνει η συνάντηση με τη Λετωνική Προεδρία που αν δεν απατώμε θα μας δώσει και μια απάντηση για το κατά πόσο θα ξεκινήσουν ξανά οι τριμερείς διάλογοι ή αν αρνούνται να ξαναρχίσουν τις εργασίες από πλευράς Συμβουλίου. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Ας δούμε καταρχάς ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και μετά θα προχωρήσουμε. Και μετά θα πρέπει να συμφωνήσουμε κι εμείς τι θα κάνουμε περαιτέρω για να ξεκινήσουν ξανά οι τριμερείς διάλογοι. Και για να φτάσουμε σε μία θέση, όπως είπε ο κύριος Βίλεν, ότι Φερρυπίν, ας πούμε, δεν έχουμε περιθώριο ευελιξίας. Μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό. Θα το δούμε ξανά. Θα το ξανασυζητήσουμε στην ομάδα αφού συναντηθείτε κύριε Χαουρέγγι με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Συζητήστε με τον πρόεδρο, συζητήστε με τους σκιώδεις και θα δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Και εγώ το ίδιο θα κάνω, ο κύριος Βίγλαν. Um με συγχωρείτε. Να με καταλάβετε καλά. Εγώ καλωσορίζω την ευελιξία. Αλλά είπα ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές επί των οποίων δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Και αν είναι να έχουμε κακό αποτέλεσμα, καλύτερα να μην έχουμε κανένα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η θέση είναι σαφής και μπορούμε να στη συμμεριστούμε. Εγώ επέμεινα στην πολιτική σημασία, στην βαθιά δημοκρατική φύση αυτής της λειτουργίας για ένα κοινοβούλιο. Οπότε, βεβαίως θα έχουμε κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτές διατυπώσεις. Αυτή η δουλειά είναι ακόμη μπροστά μας. Πρέπει να την κάνουμε, όπως είπε ο Πρόεδρος. Στον κύριο Σόλτς να πω ότι ένας καλός κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στο σώμα μας μία δραστηριότητα ερευνητική πιο συχνή. για να καταλήγουμε σε πολιτικά πορίσματα για θέματα που δεν είναι φυσιολογικά, όπου έχουν υπάρξει δυσλειτουργίες ε, αξιοσημείωτες στη συμπεριφορά ενός κράτους, μέλους και κτλ. Κάθε μέρα μαθαίνουμε πράγματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το σώμα μας σε δημιουργία τέτοιων ε, ερευνητικών επιτροπών που δεν πρέπει αναγκαστικά να καταλήξουν λέγοντα ότι αυτό φταίει, γιατί το σώμα μα δεν, δεν θέλει να αποδίδει ευθύνε. Θέλει να καταλήγει σε πολιτικά συμπεράσματα για κακή λειτουργία τη Ένωση των κρατών μελών. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Υπάρχουν σημεία από τον οποίο είμαι θα ανυποχώρητη, αλλά πρέπει να επιχειρήσουμε να καταλήξουμε συμφωνία, Αλλιώ θα είναι αποτυχία για όλου μα αν δεν το επιτύχουμε. Για όλου μα, για όλη την Ένωση. Και Πιστεύω ότι θα ήταν καλό με πορίσματα αυτού του κοινού μας διαλόγου, βεβαίως. Βεβαίως. Με τους εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων και με την πρόεδρο και εγώ ίδιος θα διεξαγάγουμε αυτή τη διαπραγμάτευση για να δούμε εάν θα καταστεί δυνατόν να προτείνουμε στο κοινοβούλιο μας μία έγκριση για να επαναλαμβάνω, έχει το κοινοβούλιο μας μία αυτονόητα, αυτονόητη δημοκρατική λειτουργία. Περιμένουμε τη συζήτηση του κύριου Χαουρέγγι και εγώ θα συναντηθώ με, τους, ε, με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και ενδεχομένως τη νομική υπηρεσία για να διευκρινίσουμε τα πράγματα και να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Τελείωσε αυτό το θέμα, να κλείσει αυτό το σημείο για να συναντήσουμε τώρα τον Επίτροπο Τίμερμανς, ο οποίος δεν έχει φτάσει ακόμα. Μπορείτε να δείτε αν έχει φτάσει. Ελπίζω να παραμείνετε στην αίθουσα, κάποιος τουλάχιστον να μείνει στην αίθουσα για τη συνάντηση αυτή. Ας περιμένουμε τον Επίτροπο. Να διατρέξουμε και τα διάφορα στο μεταξύ όμως. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και θα υπάρξουν κάποιες προτάσεις από μένα μετά τη συνάντηση με τον κύριο Τίμερμανς. Θα σας ενημερώσω και για τα όσα είπαμε με τους συντονιστές, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά αυτά θα τα δούμε μετά τη συνάντηση με τον κύριο Τίμερμαντς.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 Πρέπει να χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου, συνάδελφοι. Κάντε φασαρία. I would like to welcome uh, Vice President. Καλωσορίζω τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς ε, Τίμερμαντς. Δεν τον βλέπουμε για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε και είμαστε ευγνώμονες που έρχεστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι πρώτη φορά. Ε, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Τι άποψη έχετε για τη διαθεσμική συμφωνία και την καλύτερη νομοθεσία. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Είναι δύσκολη διαδικασία. Εμπλέκονται πολλά θεσμικά όργανα, καθώς και διάφοροι φορείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διάφορα, όργανα και σώματα, εν θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθούμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σα, Πρόεδρε, λέει ο επίτροπο, Χθε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έκανα κάτι επαναστατικό και δούλεψε. Είπα ότι δεν θα κάνω καμία εισαγωγή και θα περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Εάν συμφωνείτε κι εσείς, θα έχετε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις. Να σας δώσω λοιπόν εσάς το λόγο, να ακούσω τις ερωτήσεις σας και συνεχεία να απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές. Ε, ούτως ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτά που εσεί θεωρείτε σημαντικά. Καλή η πρόκληση. Α δώσω το λόγο καταρχά στου συντονιστέ για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Yeah. είσαι έτοιμο. Ποτέ θα είμαι πιο έτοιμο ούτω ή άλλω, Πρόεδρε, επομένω, γιατί όχι τώρα. Αρχίζω να σκέφτομαι τι μπορώ να σας ρωτήσω. Ε, κοιτάξτε, είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε την εισαγωγή και μετά να μας έρχονται και κάποιες ιδέες. Φυσικά το θέμα με απασχολεί, ε, το, βασικό θέμα και εντάσσεται στο θέμα της καλύτερης νομοθεσίας, στο το πλαίσιο της καλύτερης νομοθεσίας. Και αυτό ποιο είναι. Πώς βλέπουμε αυτή τη χρονική στιγμή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Το συζητήσαμε αρκετές φορές σήμερα. να ρωτήσω όμως και μια πιο θεωρητική ερώτηση. Ποιος νόμος είναι καλός νόμος. Τι χαρακτηριστικά έχει, πώς τον ορίζετε. Κοιτάξτε, κοιτάζετε στην πράξη πώς λειτουργεί στα κράτη-μέλη. Ανατρέχετε στο παρελθόν, ας πούμε, ε, το τι έχει κάνει η Επιτροπή. Πότε λέμε ότι είναι κακός ο νόμος θα τον πετάξουμε ή είναι καλός και άρα θα φτιάξουμε και άλλους νόμους που να σέβονται τα ίδια κριτήρια. Έτσι, εν θερμό αυτή η ερώτηση μου ήρθε. Richard, no, uh, Ο Ρίτσαρτ πρώτος. Ο Ρίτσαρτ και η κυρία Μπρέσο διαγωνίζονται για το ποιος θα πάρει πρώτο το μικρόφωνο. Ο Ρίτσαρντ, χαίρομαι που είστε εδώ. Η Κομισιόν απογοητεύτηκε φρικτά που την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να υιοθετήσει το ψήφισμα για το πρόγραμμα εργασίας του. Σημείωσα ότι δύο ή τρεις τροπολογίες είχαν την πλειοψηφία, παρότι τελικά δεν πέρασε κανένα ψήφισμα ε, δεν υπήρξε ψήφισμα για να ενταχθούν σε αυτό. Αλλά μια και είχαν την πλειοψηφία αυτές τις τροπολογίες, μπορώ να θεωρήσω ότι η Κομισιόν σημείωσε τις απόψεις που εκφράστηκαν σε αυτές τις τροπολογίες. Τροπολογίες που είχαν μια αγαστή πλειοψηφία, παρότι δεν εντάχθηκαν σε κανένα ψήφισμα. Νομίζω ότι σας εξέπληξα. Ελπίζω να μην σας ε, κατέλαβα εξαπίνης. Δεύτερη ερώτηση. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Πάντα ήμουν σκεπτικιστή για αυτή την πρωτοβουλία. Το ομολογώ. Ότι χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αν κάτι είναι καλό, αν υπάρχει μια καλή ιδέα, τότε θα πρέπει με μια απλή επιστολή στον πρόεδρο να ξεκινήσει κάτι. Μήπως πρέπει λοιπόν να καταργήσουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία τις νομικές προϋποθέσεις, τη χαρτούρα και απλούστατα. Να έχουμε μια δήλωση από την Επιτροπή ότι είναι διατεθειμένη να εξετάζει οποιαδήποτε αίτηση χωρίς να υπάρχει μια διαδικασία επαλήθευσης για κάθε υπογραφή, χωρίς να υπάρχει καταμέτρηση του αριθμού των υπογραφών. Γιατί ακόμα κι αν κάτι είναι κοντά στο ένα εκατομμύριο και κάτω από αυτό βέβαια, ε, κάποια συνέχεια πρέπει να του δοθεί, έτσι δεν είναι. Και παράλληλα γλιτώνουμε και πολύ κόπο. Η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση, πλευράς μου. για ένα σημείο κλειδί των αρμοδιοτήτων σας που είναι το better regulation, η καλύτερη νομοθεσία. Ας βγάλω τα ακουστικά με το μεταξύ, γιατί γίνεται μικροφωνισμός. Και η σχέση μεταξύ επικουρικότητας και αναλογικότητας. Μιλάμε συνέχεια για επικουρικότητα εδώ. Και τη διακρίνουμε ή μάλλον κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποτίθεται περιορισμένες και άλλες αρμοδιότητες όπου η Ένωση βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας και με βάση αυτή την αρχή καθορίζει πόσο θα παρέμβει, σε ποιο επίπεδο θα παρέμβει. παρέμβει. Και μήπως ενδεχομένως η δράση θα πρέπει να λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, στην πραγματικότητα δεν πρέπει να μιλάμε για επικουρικότητα, αλλά για αναλογικότητα. Δηλαδή για την καλή νομοθεσία, η οποία μας εξασφαλίζει καλούς νόμους, έτσι, και που αφήνει στο εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο ανάλογα με το σύνταγμα της κάθε χώρας το καθήκον να νομοθετήσουν πιο λεπτομερώς με βάση τις αρμοδιότητες αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Αυτό κινδυνεύει να περιορίσει τη δυνατότητα ελέγχου και των κρατών και της Επιτροπής των Περιφερειών και σε μικρότερο βαθμό των περιφερειακών κυβερνήσεων σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Γιατί η παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας δεν θεωρείται παραβίαση αυτή καθεαυτή. Κι όμως είναι παραβίαση. Γιατί ο πραγματικός περιορισμός της άσκησης μιας ε, αρμοδιότητας είναι απορρέει μάλλον από τις νομικές παραδόσεις και τις άλλες υπόλοιπες ας πούμε παραδόσεις, τις ιδιαιτερότητες ας πούμε που έχουν τα κράτη-μέλη. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Κάτι την άποψή μου, η αναλογικότητα είναι μία από τις βασικές πτυχές της επικουρικότητας. Ενώ πολύ συχνά τη θεωρούμε κάτι τελείως διαφορετικό, χωριστό από την επικουρικότητα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερο ερώτημα. Σήμερα το πρωί κάναμε μία συνάντηση με τους νέους της Ευρώπης. Μια ακρόαση. Δεν ξέρω κατά πόσον οι νέοι που ήταν εδώ εκπροσωπούν τη νεολαία της Ευρώπης, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Και μας είπαν δύο πράγματα. Ότι θα ήθελαν έναν εκλογικό νόμο κοινό. Για τις ευρωπαϊκές εκλογές προφανώς. Και θα ήθελαν στις ευρωπαϊκές εκλογές να ψηφίζουν και οι νέοι από τα 16 και μετά χρόνια. Φυσικά αυτό ισχύει μόνο αν υπάρχει κοινό εκλογικό νόμο. Εμεί ε, θα κάνουμε και σχετική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν τι άποψη έχει για τη δυνατότητα να ομογενοποιήσουμε τους εκλογικούς νόμους που ισχύουν ε, στα κράτη-μέλη για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Επίσης οι νέοι μας είπαν και κάτι άλλο, ακόμα πιο λεπτό και ευαίσθητο. Μας είπαν ότι πιστεύουν ότι μια και οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν την Ευρώπη και για να την καταλάβουν η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ένα απλό συνταγματικό κείμενο με λίγα άρθρα που θα μιλάει για τις ε, βασικές γενικές αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρώπη ούτως ώστε να καταλαβαίνουν οι πολίτε και κυρίως οι νέοι πολίτες πώς λειτουργεί η Ευρώπη, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο μια σειρά από νόμους, νομοθετήματα, κανονισμούς, οδηγίες που είναι καλοφτιαγμένα μεν, αλλά δύσκολα και τεχνικά. Αυτά τα λέω έχοντας υπόψη το μέλλον της Ευρώπης. Είναι δύσκολη αυτή η στιγμή, γιατί δεχόμαστε επιθέσεις στις αρχές μας, στα πιστεύω μας, ακόμα και στην ίδια μας τη ζωή. Πιστεύετε ότι μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να ξεκινήσει. Γιατί αυτά μας τα είπαν οι νέοι πολίτες μας. Ε, και πολλοί από εμά, λιγότερο νέοι από αυτούς, θα ενδιαφερόμασταν για τέτοια θέματα και για τέτοια συζητήσεις. Ο Καλώ uh, Καλώς ήρθατε κύριε Τίμερμανς. Θα ήθελα να δω τα πράγματα ε, πιο αποστασιοποιημένα. Ε, να μου πείτε τη γνώμη σας για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, στο απότερο μέλλον. Ε, πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί προς την κατεύθυνση του της ε, ε, ενιαίας ε, αντιμετώπισης ή θα, θα ακολουθήσει πιο ευέλικτους δρόμους. Ο, ο πρόεδρος Επιτροπής έλεγε ότι είναι υπέρ μιας δίκαιης λύσης του προβλήματος με το Ηνωμένο Βασίλειο. Την άλλη μεριά οι Times λένε ο, σε ένα άρθρο στην Κυριακή ότι, ε, ότι θα κατευθυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ προς την ιδέα του ότι θα είναι κάτι το ενιαίο και όποιος δεν είναι ικανοποιημένος μπορεί να, την, να, να φύγει, να την εγκαταλείψει. Εσάς ποια είναι η άποψή σας. Είναι ένα κρίσιμο θέμα η υπόσχεση του κύριου Γιούνκερ πριν την εκλογή του ε, που είχε συζητηθεί στην ομάδα μας στην ECR ε, ε, ενδεχομένως δεν αφορούσε μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και όλες οι υπόλοιπες χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Οπότε είχε δημιουργήσει ελπίδες και όχι μόνο σε χώρες αλλά και σε κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν ενδεχομένω να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με λιγότερες δεσμεύσεις από ό,τι οι υπόλοιπε. Ε, τώρα, δείχνει ο κ. Γιούνκερ να πηγαίνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Εσείς, κ. Τίμερμανς, πιστεύετε ότι θα πρέπει να τηρηθεί η παλαιότερη υπόσχεση του Προέδρου σας, ε, ο οποίος δείχνει να την προδίδει ή είσαστε στο στρατόπεδο Γιούνκερ που κατά βάση λέει όποιος του αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φύγει, να κατέβει από το τρένο. Πιστεύετε ότι κράτη και κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν αυτό ακριβώς το πράγμα μπορούν να παραμείνουν. Θα υπάρχει ε, ευελιξία. Πολύ ωραία. Ο κ. Βίλαντ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Όλοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη νομοθεσία. Αλλά ένα δίκαιο που δεν εφαρμόζεται, όσο καλό και να είναι θεωρητικά, είναι κακό. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να προσέξουμε να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή των νομοθετημάτων μας πριν δημιουργήσουμε και άλλους νόμους, πριν αποτιμήσουμε τους παλιούς Μήπως θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να δούμε εάν εφαρμόζονται οι νόμοι που έχουμε. Δεύτερον, είστε αρμόδιος, αρμόδιος για τις ε, διοργανικές σχέσεις. Θα μου άρεσε πολύ αν μαζί με τον κύριο Ατόντο που είναι εισηγητής για τις ε, επιτροπές, ε, εξεταστικές επιτροπές, αν μπορείτε να επιτύχετε περισσότερα για αυτό το θέμα. Επίσης, πάντα για τις διοργανικές σχέσεις, νομίζω ότι είναι σοβαρή κακή εξέλιξη ότι έχουμε πάνω από 90% συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης. Θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Νομίζω ότι η πολιτική κουλτούρα σε ολόκληρη την Ήπειρό μας έχει οδηγήσει σε μια πρακτική τριών αναγνώσεων που συνήθως είναι δημόσιες. Δεν είναι δυνατόν εμείς να συμφωνούμε εν κρυπτό. Αλλιώς ε, τι καταλαβαίνουμε ως κοινοβούλιο ότι κάνουμε. Κάτι άλλο που είναι και εφαρμογή δικαίου και διοργανικές σχέσεις. Θα επιθυμούσα. Δεν ξέρω αν είναι υποκειμενική εντύπωσή μου, αλλά τουλάχιστον εγώ έχω την εντύπωση και άλλοι και το βλέπω και στην Επιτροπή Αναφορών, ότι λοιπόν όταν υπάρχουν προβλήματα πολύ πιο εύκολα λαμβάνονται μέτρα κατά μικρότερων κρατών μελών σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Και ακόμη και για λεπτομέρειες αργεί πολύ η Κομισιόν. Ένα παράδειγμα. Δεν θα, δεν θα ξέρουν οι συνάδελφοι ότι στα μεγάλα αεροδρόμια υπάρχει ένα κτηνιατρικό ιατρείο. Και αυτό σημαίνει ότι επειδή ταξιδεύουν λοιπόν τα ζώα, ε, υπάρχει μετάδοση για την δροσόφυλα, τη μίγα που ζει μία μέρα μόνο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να επιτρέπουμε τέτοια, ε, τέτοιες καταστάσεις. Η Κομισιόν είπε ότι θέλει να μην ανεχθεί αυτές οι καταστάσεις. Όμως καθυστερεί. Επανειλημμένα μας έχει πει ότι θα διορθώσει αυτή την κατάσταση και δεν το έχει κάνει. Τώρα, κράτος δικαίου. Θα περίμενα από την Κομισιόν και ειδικώς από εσά πώς τα, δικαστήρια στα κράτη-μέλη απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια προκαταρκτική απόφαση και πώς αποφασίζουν εάν θα αποφασίσουν τα ίδια. Διότι με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζεται διαφορετικά το δίκαιο. Και αυτό είναι λάθος. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν περιμένω ε, εκτεταμένη απάντηση σήμερα, αλλά το θέμα είναι πώς κατανοούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με την χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι παραδοσιακά θεωρούσαμε ότι τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά η σύγχρονη αντίληψη του δικαίου με βάση τι αποφάσει του δικαστηρίου είναι ότι αν τα κράτη-μέλη δημιουργούν εθνικό δίκαιο και με βάση το εθνικό δίκαιο περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα, τότε αυτοί οι περιορισμοί αυτοί οι περιορισμοί δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί. όχι λοιπόν μόνο πρέπει να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και για το εθνικό δίκαιο δεν θα πρέπει να περιορίζεται μέσω του εθνικού δικαίου. Αυτή είναι η ε, σύγχρονη αντίληψη δικαίου. Και τελευταίο. Υπάρχει μια μικρή ομάδα εργασίας για τον κανονισμό με τον Γκόρμετ, Άντερσον και Σόλτς και προκύπτει ένα θέμα διότι έχουμε υπερβολικό αριθμό ερωτήσεων από το Κοινοβούλιο προς την Κομισιόν. Και αυτό προκαλεί πολλές ανησυχίες στην Κομισιόν. Είμαστε δεδεθειμένοι να πούμε ότι επειδή πολλές είναι απλώς ερωτήσεις για στατιστικά στοιχεία, θα είχε έννοια να παρακαλέσουμε τους συναδέλφους να μην απευθύνουν στην Κομισιόν τέτοιε ερωτήσεις, να απευθύνονται αλλού. Αλλά κύριε Τίμερμανς, σε αντιστάθμιση, θα ήθελα τότε οι απαντήσεις που μας δίνει η Κομισιόν να είναι λίγο λιγότερο κενές περιεχομένου. Δεν έχω θέσει πολλές ερωτήσεις ε, ως βουλευτής, αλλά μερικές ε, απαντήσεις ήταν ε, στο όριο της αγένειας. Δεν είναι δυνατόν όταν κάνει κανείς μια λογική ερώτηση να λαμβάνει μια τέτοια κενή απάντηση. Θα πρέπει να ανέβει το επίπεδο των απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όταν μιλούσε η κυρία Μπρέσο, έβγαλε τα ακουστικά της. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι ε, στο Μόναχο. Ο Χένρι Κίσιγκερ μιλούσε και είχε κάτι στο μυαλό του. Ή μάλλον είχε κάτι στο κεφάλι, στο κεφάλι του. Α, ακουστικά προφανώς. Τα έβγαλε κάποια στιγμή και είπε «Α, άκουγα τον εαυτό μου στα γερμανικά και αισθανόμουν πολύ γερμανο, είπε με γερμανική προφορά στα αγγλικά. Τέλο πάντων, να σα απαντήσω σε ερωτήσει σα. Θα προσπαθήσω να μην τα χρησιμοποιήσω τα ακουστικά, αλλά αν αρχίσετε να μιλάτε πολωνικά, κυρία Χιούμπνερ, θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσω. Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Τονίζω ότι πιστεύω πως αυτό το εργαλείο μπορεί να γίνει πολύ σημαντικό. Σημαντικό για πολιτικό διάλογο, για την κοινωνία. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν ε, μεγάλη ευθύνη και δεν πρέπει να, φυλακι... να φυλακίσουν τον εαυτό τους ε, στη φούσκα αυτή των Βρυξελών, στο γυάλινο πύργο των Βρυξελών. Ε, έχω αυτή την τάση, το αισθάνομαι μετά από τρεις μήνες που είμαι εδώ. Θα πρέπει να επανασυνδεθούμε με τον κόσμο. Και αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να είναι ένα καλό εργαλείο για αυτό, για αυτή την επανασύνδεση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό τον τρέχοντα κανονισμό. Θα πρέπει να τον ξαναδούμε βέβαια για να βεβαιωθούμε ότι γίνεται. Όμως, η Κομισιόν έχει την νομική υποχρέωση, αν υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία, να εξασφαλίσει ότι εντάσσεται στο σημερινό νομικό πλαίσιο που είναι η συνθήκη και οι κανονισμοί. Έχει υποχρέωση να το κάνει αυτό, να επαληθεύσει αυτό το πράγμα η Κομισιόν και αναγκαστικά θα πρέπει να σεβαστεί και τη συνθήκη και τον κανονισμό η Κομισιόν, γιατί είναι ο θεματοφύλακας αυτών. Αν όμως με αυτά τα νομικά δεδομένα και προϋποθέσεις καταλήξουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να αποτελέσει βάση για να συνεχιστεί ένας πολιτικός διάλογος με του ανθρώπου που μπήκαν στον κόπο να υπογράψουν μια τέτοια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και θα μπορούσε επίση να είναι χρήσιμη γιατί εν συνεχεία μπορούν να ενταχθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αντιδράσουν στην πρωτοβουλία αυτή και να μπουν στη συζήτηση και αυτή. Και όπω είπα και στην ακρόασή μου, η Κομισιόν θα είναι ανοιχτή να χρησιμοποιηθεί με πιο πολιτικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, να γίνει μεγαλύτερη πολιτική χρήση αυτή τη πρωτοβουλία, περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι στο παρελθόν. Αν αντιδράσουμε την πρωτοβουλία αυτή. Και η αντίδραση δεν είναι αυτό που ήθελε ο κόσμος. Δεν είμαστε εξάλλου υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε μαζί τους, έτσι. Μπορεί να είναι αρνητική η αντίδρασή μας. Μπορεί όμως και αυτή η αρνητική αντίδραση να είναι η απαρχή ενός πολιτικού διαλόγου. Και το θέμα του πολιτικού διαλόγου είναι ότι δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις στο τέλος του διαλόγου, αλλά να συμφωνήσει ότι ο διάλογος έχει νόημα να γίνει. Και ότι γίνεται αυτός ο διάλογος με σεβασμό όλων των απόψεων που ακούγονται σε αυτόν και νομίζω ότι είναι η ευθύνη μου να δείξω ότι η Κομισιόν ενεργεί με υπευθυνότητα όταν αντιμετωπίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Ο κ. Κόμπαρτ είπε ότι ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε μια ενδεχόμενη αλλαγή των κανόνων. Το είπα και εγώ στην ακροασή μου, ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να δούμε όμως πιο προσεκτικά τον κανονισμό για να δούμε αν υπάρχει περιθώριο αλλαγή. Ακόμα όμως και αν δεν τον αλλάξουμε, μπορούμε να βελτιώσουμε τον πολιτικό διάλογο βάσει τις προσπάθειες που κάνει ο κόσμος, οι πολίτες, να προχωρήσουν σε αυτή την πρωτοβουλία, σε, αυτές τις... σε αυτά τα αιτήματα, αν θέλετε. Σε αυτές τις αναφορές, για να το πούμε έτσι. Τώρα, για την ερώτηση, τι, ποιος νόμος είναι καλός. Δύσκολη ερώτηση. Ας σας δώσω κάποια στοιχεία. Ένας κανός νόμος θα πρέπει να είναι βιώσιμος. Δεν έχουμε την οικολογική βιωσιμότητα, την κοινωνική, την οικονομική βιωσιμότητα. Θα πρέπει να υπάρχει και νομική βιωσιμότητα. Έχει νόημα να ξαναδούμε το νομοθετικό σώμα που έχουμε και να δούμε αν είναι βιώσιμο. Και αμέσως εδώ μπαίνει ένα πρόβλημα για εμάς τους πολιτικούς. Όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο κράτος μέλος. Οι πολιτικοί θέλουν τους νέους νόμους, θέλουν να φτιάχνουν νέους νόμους, αλλά είμαστε καταστροφικοί στην αναθεώρηση των δικών μας παλιών νόμων. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εξετάζουμε και αν το νομοθετικό μας σώμα που δημιουργήθηκε στο παρελθόν εξακολουθεί να είναι σημαντικό σήμερα, ε, να είναι βιώσιμο σήμερα. Ένα πρόγραμμα refit θα πρέπει να εξετάζει λοιπόν και την ισχύουσα νομοθεσία. Και ένα άλλο, μια άλλη απάντηση για το ποιο νόμο είναι καλό. Πρέπει να δούμε πώς δημιουργείται η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αρχίζουμε την νομοθετική διαδικασία στην Κομισιόν, κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου του νέου, της νέας νομοθεσίας. Είναι ευθύνη των υπηρεσιών της Κομισιόν να την κάνουν. Αν γίνει αυτή η μελέτη, το αποτέλεσμα υποβάλλεται στο Συμβούλιο Εξέτασης των Μελετών Αντιχτύπου και 40% των μελετών αυτών στέλνονται πίσω γιατί δεν αρέσουν στο Συμβούλιο και θα πρέπει να ξανασυνταχθούν. Επομένως πρέπει να υπάρχει, να είναι υψηλό το επίπεδο του, της νέας νομοθεσίας, του νέου νομοθετήματος για να προχωρήσει. Ας ξαναδούμε λίγο την νομοθετική διαδικασία. Ακόμα και αν έχουμε συντάξει ένα άλογο στην αρχή της διαδικασίας, συχνά το αποτέλεσμα είναι μια καμήλα. Γιατί το διαπραγματευόμαστε στο συμβούλιο, με το Συμβούλιο. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη και δεδομένη τη ε, περιπλοκότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, με τόσε πολλέ ε, διαφορετικέ απόψει, πολιτικέ πραγματικότητε, μερικέ φορέ επικεντρωνόμαστε στο να πετύχουμε τη την ε, συμφωνία και ξεχνάμε το αν η συμφωνία είναι σαφής. Αν θα έχει επίπτωση, την προσδοκόμενη επίπτωση, εν στα κράτη-μέλη που θα την εφαρμόσουν. Συχνά αυτή η σκέψη, το, το τι επίπτωση θα έχει, είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την ανάγκη να πετύχουμε τη συμφωνία. Θέλουμε γρήγορη συμφωνία και δεν ελέγχουμε την ποιότητα. Αν θέλουμε λοιπόν να φτιάχνουμε καλούς νόμους στο μέλλον, θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους τα τρία εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα μοιράζονται την ευθύνη για την μελέτη αντικτύπου του τελικού προϊόντος, πριν εφαρμοστεί δηλαδή στα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν ιδανικά η καλύτερη στιγμή, θα ήταν η καλύτερη στιγμή για να κρίνουμε το νομοθέτημα, που είναι το αποτέλεσμα της λογικής μας προσπάθειας. Για να ξέρουμε αν, ας πούμε, αυτό που φτιάχνουμε είναι αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε αρχικά. Αυτό που προκύπτει, εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο στοιχείο του καλού νόμου είναι ότι δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώριο για πολλαπλέ ερμηνείε. Τεράστιο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μα και λόγω αυτή τη ποικιλομορφία έχουμε τάση να προτιμούμε αρκετά εύκολα την οδηγία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο κανονισμός είναι πολύ πιο άκαμπτος στο τι ερμηνείες επιδέχεται. Γι' αυτό προτιμούμε τι οδηγίε, οι οποίε θα πρέπει να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία, να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία. Και αν η οδηγία δεν είναι σαφή στο, ως το τι θα πρέπει να ενσωματώσει το κράτο μέλο, υπάρχει κίνδυνο κανονιστικού υπερθεματισμού από τα κράτη-μέλη. Και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια κατά κόρον αυτό το πράγμα. Ο κανονικός, κανονιστικός υπερθεματισμός. Ένας καλός νόμος είναι ένας νόμος που δεν χρειάζεται τα κράτη-μέλη να πάνε πέραν αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι πάρα πολύ ποικιλόμορφη για να μπορέσει να πει ναι, τέρμα οι οδηγίες, ας πάμε στους κανονισμούς. Είμαστε υπερβολικά διαφορετικοί. Και υπάρχουν και διαφορές ακόμα και εντός των κρατών μελών. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη τόσο συγκεντρωτικά όσο το Λουξεμβούργο ή η Ολλανδία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την εσωτερική δομή των κρατών μελών και τι διαφορετικέ πραγματικότητες και την ποικιλομορφία στο εσωτερικό του κάθε κρατου μέλου. Επίση, πρέπει να είμαστε πολύ πιο ακριβείς για να παρεμποδίσουμε τον κανονιστικό υπερθεματισμό στα κράτη-μέλη και να μην δίνουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να λένε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Νομοθέτημα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Μπρέσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η επικουρικότητα και τι είναι η αναλογικότητα σε νομικό επίπεδο. Εγώ ήμουν πολιτικό σε εθνικό επίπεδο αρχικά και ξέρω πολύ καλά ότι πολύ συχνά αυτό που παρουσιάζεται ως αρνητικός έλεγχος επικουρικότητας είναι μια αρνητική γνωμοδότηση για το περιεχόμενο ενός νομοθετήματος. Νομίζω ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν απόλυτο δικαίωμα να έχουν αρνητική γνώμη για το περιεχόμενο του νομοθετήματος, αλλά θα πρέπει να δικαιολογούν αυτή την αρνητική γνώμη στους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Εάν θέλουμε το σύστημα να αποτελεσματικό, η αναλογικότητα θα πρέπει να είναι αν υπάρχει νομική, να εξετάζουμε το αν υπάρχει νομική βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δράσει. Και ο δεύτερος έλεγχος είναι αν το μέσον που θέλει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανάλογο ως προς τον επιδιεκόμενο στόχο. Και εδώ υπάρχουν διαφορές ως προς τα κράτη-μέλη. Αν έχεις υψηλό, υψηλά συγκεντρωτικό συγγνώμη, πολύ συγκεντρωτικό ένα κράτος μέλος, ε, έχεις άλλη γνώμη συνήθως από ότι ένα κράτος το οποίο είναι όπως η Ιταλία, η Γερμανία κτλ. Επομένως, η αναλογικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αν το κάνουμε σωστά όλο αυτό και αν υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων αλλά και των εθνικών κοινοβουλίων και του ευρωπαϊκού και υπάρχει και θετική στάση, νομίζω ότι μπορούμε τότε να φτιάξουμε καλύτερου νόμου. Αλλά ας μην είμαστε αφελείς. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι μερικές φορές αυτό που παρουσιάζεται ως έλεγχος επικουρικότητας είναι ότι ένα εθνικό κοινοβούλιο λέει απλούστατα «Α, δεν μας αρέσει αυτό το νομοθέτημα, δεν μας αρέσει το περιεχόμενό του». Εντάξει, καλό και αυτό, αλλά τότε θα πρέπει να το πεις αυτό στους εκπροσώπους του Συμβούλιο, οι οποίοι διαπραγματεύονται αυτό το νομοθέτημα. Να μην λέτε, να μην λένε αυτοί οι εκπρόσωποι λέει, το Εθνικό Κοινοβούλιο στην Κομισιόν, α, δεν μας αρέσει αυτό το νομοθέτημα γιατί δεν είναι αναλογικό ας πούμε και δεν έχει ελεγχθεί η αναλογικότητά του. Όχι. ιδέα ενός κοινού εκλογικού νόμου ή ενός κοινού εκλογικού συστήματος. Δύσκολο θα είναι αυτό. Δεδομένων των πολλών διαφορών που υπάρχουν στην εκλογική νομοθεσία των κρατών μελών. Εντάξει, λογικά στέκει αυτό που λέτε, αλλά πολιτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό και αν το δεχθούν τα κρατη Ας μην τρέφουμε τέτοιες φρούδες ελπίδες. Ο κ. Κόμπετ είπε ότι δεν υιοθετήθηκε ψήφισμα για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Σωστό. Μπορούμε να πούμε πολιτικά εντάξει τότε, συνεχίζουμε αυτά που προτείναμε. Εγώ θα προτιμούσα όμως να μας είχε δώσει κάποια έτσι, κάποιο ψανατολισμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί τότε η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας είχε φωτίσει λιγάκι ως προς το τι επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Πλειοψηφικά πάντα, έτσι. Είναι κρίμα που δεν έγινε κάτι τέτοιο. Είναι κρίμα για τις διαθεσμικές μας σχέσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε και υποχρεωμένοι ως Κομισιόν να δούμε όλα τα ψηφίσματα που περάσατε εσείς, να τα συγκρίνουμε και να βρούμε τον κοινό παρανομαστή τους. Εγώ θα έλεγα, εσείς έχετε τον μπαλάκι. Φτιάξτε ένα ψήφισμα, βρείτε πλειοψηφία και τότε η Κομισιόν θα το λάβει υπόψη το ψήφισμα αυτό. Δεν μπορείτε να μας ζητάτε εμάς να αρχίσουμε να κάνουμε copy-paste, ας πούμε, των διαφόρων ψηφισμάτων που έχετε περάσει για το πρόγραμμα εργασία μας. Εντάξει, μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες, αλλά δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Α, για τις τροπολογίες θέλετε να μιλήσω. Τις εγκεκριμένε τροπολογίες, μόνο για αυτές. Οκ. Τι είναι η Ευρώπη. um... Πόσο χρόνο έχουμε. I think this is... Η κυρία Μπρέσο αναφέρθηκε στους νέους και νομίζω ότι οι νέοι θέτουν το ίδιο ερώτημα που θέτει ο κύριος ε, Μέσσερ Σμιτ και ενδεχομένως και ο κύριος Βίλαντ εν μέρη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στους τρεις. Κατ' εμέ, η Ευρώπη είναι ένα μέρος όπου δεν γίνεται συζήτηση για το ποιο ανήκει σε αυτήν την Ήπειρο. Η Ευρώπη είναι μια περιοχή ε, όπου ορισμένοι μειοψηφίε δεν φοβούνται για το μέλλον τους. Μπορεί να συζητάμε για τις δομές, για τα όργανα, για, τα, για την βελτίωση νομοθεσίας, αλλά 70 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ε, μία από τις κοινότητες που ε, είναι κρίσιμες για την ιστορία όλων, ε, αρχίζει και ανησυχεί για τη θέση της στην Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως είναι μια περιοχή του κόσμου όπου ισχύει το κράτος του δικαίου, όπου οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τα κράτη-μέλη ε, μας εμποδίζουν στο να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Αν δείτε την κοινή αγορά, το ευρώ, όλα όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 60 χρόνια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όλα ε, έχουν ως ε, στόχο να δημιουργηθεί ένας χώρος ελευθερίας κράτους δικαίου, ε, ελευθερίας ε, πίστης, ε, ελευθερίας έκφρασης κλπ. Αυτά είναι η Ευρώπη. Αν με ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό για τα κράτη-μέλη, να σας πω το εξή. Οι συνθήκε τη είναι σαφείς. Αν αυτή η οικοδόμηση της Ευρώπης δεν ικανοποιεί κάποιον, είναι ελεύθερος να φύγει να εγκαταλείψει αυτή την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αλλά πιστεύω, και δεν είναι μόνο η προσωπική μου άποψη, είναι και άποψη όλη τη Κομισιόν και του Προέδρου τη, ότι αν υπάρχουν ανησυχίε για το πώ λειτουργεί και διαρθρώνεται η Ευρώπη σήμερα, και είμαι σίγουρο ότι όλοι μας έχουμε προβλήματα και επιφυλάξει σε σχέση με το πώ εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μα, ανεξαιρέτω, αν υπάρχουν θα πρέπει να ακούσουμε αυτές τις ανησυχίες προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέποντας ε, την ευρύτητα του φάσματος των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλαβαίνει κανείς ότι οι ψηφοφόροι ε, είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφοι ε, στις απόψεις τους, ιδεολογίες τους κλπ. Θα πρέπει να ακούσουμε όλες αυτές τις φωνές. Αλλά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνεργασία βασίζεται σε μια σειρά αρχών, βασίζεται σε κάποιες συνθήκες και αυτό έχει βοηθήσει την Ήπειρό μας να αναπτυχθεί για πολλές δεκαετίες ειρηνικά και νομίζω ότι είναι βιώσιμο και στο μέλλον. Κάποιοι στο, κάποιος Βασίλειο είχε πει, ένας πρώην Πρωθυπουργός νομίζω, ότι δεν θα χάνε τον ύπνο του αν, η, το Βασίλειο έφευγε ή κατέβαινε από το τρένο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εγώ νομίζω κάτι τέτοιο θα ήταν τραγικό για το Ηνωμένο Βασίλειο, αν εγκατέλειπε την Ευρωπαϊκή Ένωση Βέβαια, αυτό είναι μια απόφαση που θα την ε, λάβει ο, ο λαός στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, ο οποίο είναι κυριαρχό. Όμως, η ε, λογική λέει ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μια αγορά 500 εκατομμύριων ε, πολιτών θα είναι σίγουρα καλύτερη από ό,τι εκτός. Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο λαός. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι η Κομισιόν θα, κάνει, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αισθανθεί βολικά, άνετα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γνωρίζω, γιατί το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο της Κομισιόν, ότι ο κ. Γιούνκερ έχει την ίδια άποψη. Δεν ξέρω τι είπε ακριβώ το Παρίσι, αλλά να σας πω εγώ μερικά μου λόγια. Πάντα υπάρχουν και κάποια όρια στο περιθώριο ελιγμών που διαθέτουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε την αλφα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει φύση. Η συνεργασία που βασίζεται πάνω στις αρχές της συνθήκης είναι ο κανόνας. Όλοι σεβόμαστε τη συνθήκη, ακόμα και οι πιο ισχυρές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αφαιρέσουμε αυτή τη συνθήκη, δεν μπορεί να σταθεί το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το όριο, νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα διαρθρωθεί η Ευρώπη στο μέλλον. Αυτό είναι δυνατόν. Και πιστεύω φανατικά ότι ο σεβασμός των θεμελιών δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, η, η διάρθρωση γύρω από τους όρους και τις αρχές ε, μιας συνθήκης είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επόμενες δεκαετίες. Τώρα, αν θέλουμε βελτίωση της νομοθεσίας, ναι, θα πρέπει να δούμε και το θέμα της εφαρμογής. Και η Κομισιόν είναι υπεύθυνη να ε, εγγυάται ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εφαρμόζεται όπως πρέπει να εφαρμοστεί. Και αν αυτό δεν συμβαίνει, η Κομισιόν έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ε, κινεί προσφυγές, διαδικασίες ε, Ε, που να υποχρεώνουν τι χώρε να συμμορφωθούν. Τώρα, αν ο κ. Βίλαν θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με τη Γερμανία, <laughs> μπορεί. Αν έχετε να μου πείτε συγκεκριμένα στοιχεία, εγώ δεν το πιστεύω βέβαια. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Κύριε Βίλαντ, ο κ. Βίλαντ εξέφρασε ε, ανησυχίες, γιατί είπε ότι η Κομισιόν ε, είναι πιο αυστηρή με τα μικρά κράτη-μέλη παρά με τα μεγάλα. Οπότε είπα θα το ξαναδούμε πιο κοντά, να δούμε αν είμαστε υπερβολικά επίοικείς με τη Γερμανία. Εγώ δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, είναι δίκαιη στην προσέγγιση, σας, της. Ακόμα και όταν δεν ήμουν μέλος της Κομισιόν δεν είχα τέτοιου είδους παράπονα. Δεν θεωρούσα ότι η Κομισιόν είναι αδική ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έκανε λάθος με το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη όταν αρχικά ήταν πολύ αυστηρή με την Πορτογαλία. Και ε, λίγο αργότερα ε, δέχτηκε ότι η Γερμανία και η Γαλλία δεν θα πρέπει να έχει την ίδια αυστηρή μεταχείριση. Αυτό ήταν λάθο και δεν πρέπει να το επαναλάβουμε. Οι ίδιοι κανόνε θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλου, μικρού και μεγάλου. Να δω τι υπόλοιπε ερωτήσει. Για το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη θέση του δικαστηρίου. Ε, η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, από όσο γνωρίζω, δεν επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μόνο, μόνο αλλά και τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι, αυτή νομίζω η κατάσταση. Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ασφαλώς, ναι. Και μια και μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ε, να σας πω ότι εξετάζουμε προσεκτικά τη γνώμη του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και η Επιτροπή θα λάβει θέση μόλις τελειώσει η αξιολόγηση. Αλλά να σας πω ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ενταχθεί στην ε, ε, ε των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε, πρόεδρος, έχουμε ακόμα οκτώ συναδέλφους ε, από ένα λεπτό στον καθένα για να δώσουμε και λίγο χρόνο στον Επίτροπο, για να δώσουμε και πέντε λεπτά στον Επίτροπο. Οπότε ένα λεπτό κατάτομο. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι τα εθνικά κοινοβούλια κάνουν κατάχρηση της αρχής της επικουρικότητας και έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπη όταν δίνει τη νομική βάση για κάποια νομοθετήματα καταχράται της αρχής επικουρικότητας και δίνει πολύ γενικόλογες αιτιολογήσεις και επιχειρήματα για το πώς πρέπει να ασκηθεί η αρχή της επικουρικότητας. Αλλά συγκεκριμένα για κάποιες πρακτικές που είναι κατά της ε, λειτουργίας της ε, ελεύθερης αγοράς. Η γερμανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, έκανε κάποιες ανακοινώσεις για τις ε, ξένες εταιρείε μεταφορών ότι πρέπει να εφαρμόζουν το, τη γερμανική νομοθεσία για τις ελάχιστες απολαβές. Ε, πώς αποτιμάτε αυτές τις πρακτικές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάινεν, ε, αγαπητέ Φραντς, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρώτη Αντιπρόεδρε, για μας εκπροσωπείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλά θέματα, όχι μόνο για καλύτερες ε, κανονιστικές διατάξεις, ευρωπαϊκές αξίες, κράτος δικαίου, εξέλιξη της Ένωσης. Το ερώτημα είναι εάν θα έχουμε μία νέα προσέγγιση για την ε, αξία που έχει η Ένωση, για ποιο λόγο ύπαρξης έχει η Ένωση, ποιες είναι οι αξίες της και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ε, ευρωσκεπτικισμό. Είχαμε προηγουμένως την κυρία Βάλστρομ, ε, μετά την κυρία Ρέντινγκ. Τώρα είστε εσείς που μαζί μας προσπαθεί να οργανώσει την κοινή μας αντιμετώπιση. Και το ερώτημα είναι τι επίκειται λοιπόν. Δεύτερον, καλύτερες κανονιστικές διατάξεις. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε δημιουργήσει την εντύπωση ότι η εθνική νόμοι είναι υψηλού πολιτικού επίπεδου, ενώ η ευρωπαϊκή νόμοι είναι τρομερή γραφειοκρατία. Εντάξει, ορισμένες φορές είμαστε κάπως ασαφείς και ίσως μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Ξέρω από τους προέδρους του δικαστηρίου του δικού μας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι πολλές φορές είναι σχεδόν ανεφάρμοστοι γιατί υπάρχουν πολλές ασάφειες. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ορισμένα δεν είναι τόσο καλά. Τρίτον, για τα εθνικά κοινοβούλια λυπάμαι ιδιαίτερα που η κίτρινη κάρτα φέρνει τα κοινοβούλια σε αμυντική θέση. Πρέπει να πούνε τι δεν είναι καλό, ενώ η δική μας πρόθεση ήταν να συμπεριληφθούν σε μια συζήτηση που θα λέει τι θέλουν, τι θεωρούν ότι είναι σκόπιμο για να διαμορφώσουμε ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια μία, ένα θετικό θεματολόγιο. Α, η Μάιτε θέλει. Ο κύριος Κατρούγαλος. Ευχαριστώ. Ακούσατε, άκουσα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη δέσμευσή σας για να ξεκινήσουμε ένα διάλογο. Δύο σύντομες ερωτήσεις, αλλά θέλω παρακαλώ πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Την Κυριακή έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα. Και κατά πάσα πιθανότητα η νέα κυβέρνηση θα έχει πολύ διαφορετική εντολή από την προηγούμενη. Γιατί κεντρικό σημείο του προγράμματός της είναι η αναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων. Ερώτηση λοιπόν. Εσείς ως Επιτροπή και προσωπικά θέλετε να συμμετάσχετε σε έναν διάλογο με τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Εάν η νέα κυβέρνηση θέλει αναδιαπραγμάτευση εντός του πλαισίου του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου. Γιατί άκουσα από επιτρόπους το επιχείρημα ότι πάκτα sunt servanta και ότι η αλληλεγγύη εξαρτάται από την τήρηση των συμπεφωνημένων. Και θα ήθελα τη γνώμη σας. Ισχύει αυτό. Γιατί γίνονται εκλογέ τότε. Γιατί χρειάζεται να ψηφίζουμε. Γιατί χρειάζεται να έχουμε δημοκρατία. Εάν ένας λαός κυρίαρχα δεν μπορεί να αλλάξει. Επαναλαμβάνω όχι επί των συντακτικών ε, στοιχείων, αλλά επί ορισμένων σημείων της ε, πολιτικής και των επιλογών πολιτικής. Και δεύτερον, εάν ε, θέλετε να γίνει αναδιαπραγμάτευση θα την κάνει η Τρόικα, ένα άτυπο όργανο ή είστε διατεθειμένοι η αναδιαπραγμάτευση να γίνει εντός των οργάνων της Ένωσης και ιδιαίτερα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάουλου Ραντζέο. Πολύ σύντομα γιατί έχει τεθεί και έχει απαντηθεί μάλιστα η ερώτηση. Έχει να κάνει με την ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. και την ένταξη χωρών και τη γνώμη του δικαστηρίου. Θέλω να πω λοιπόν ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι είναι αποφασισμένη η Επιτροπή να εφαρμόσει τις συνθήκες. Και έχει την πολιτική βούληση να συνεχιστεί η διαδικασία για την προσχώρηση της Ένωσης στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστάλντο. Καλησπέρα, Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ας μιλήσω Ιταλικά, μια και είσαστε λάτρης των ε, Ιταλικών και έχουμε και την ίδια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Α, τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε, την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά τις διαθεσμικές σχέσεις στην πραγματικότητα θέλω να πάρετε μια δέσμευση. Όχι να σας κάνω ερώτημα. Θέλω να συμμετέχουν περισσότερο όλες οι πολιτικές ομάδες στα διάφορα όργανα. Να σας δώσω ένα ε, συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί εγώ ανήκω και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ εξαρτάται και από την Ειδική Επιτροπή, που αντιστοιχεί λιγάκι σε αυτό που υπάρχει και στην, στο στην Ιταλική πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι μια επιτροπή που έχει ε, στην κατοχή της λεπτές και ευαίσθητες πληροφορίες. Αποτελείται από πέντε μέλη. Χρησιμοποιούν τη μέθοδο DON'T για να, για να διοριστούν, ας πούμε. Και οι τρεις είναι από το ΕΛΚ και οι δύο από τους σοσιαλιστές. και η ECR πήρε τη θέση του Άλντε, των φιλελεύθερων δηλαδή, μετά τις εκλογές. Πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουμε συνθέσεις πιο αντιπροσωπευτικές των, της ετοιμιγορίας των πολιτών. Γιατί έτσι δημιουργούνται δύο κατηγορίες ευρωβουλευτών κατηγορία Α και κατηγορία Β και δεν νομίζω ότι θέλουμε κάτι τέτοιο στις εργασίες μας. Ελπίζω να γίνει πραγματικός διάλογος, επικοδομητικός μαζί σας, εδώ σε αυτή την Επιτροπή, για να βρούμε λύσεις εναλλακτικέ σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη μέθοδο DON'T. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Κύριε Αντιπρόεδρο, χαίρομαι πολύ που ο κύριος Στόιμπερ είναι ειδικό σύμβουλος τώρα και προσβλέπω στην συνέχιση της πολύ καλής εργασίας του για καλύτερες κανονιστικές διατάξεις. Για τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμενους όμως χρειάζεται κάποια διευκρίνηση για να δούμε ακριβώς πώς θα αποτιμήσουν την επίπτωση της νομοθεσίας. Δεύτερον, πολύ ενδιαφέρουσα την προσπάθεια μεταγραφής του κεκτημένου. Οι χώρες που θέλουν να ενταχθούν διαπραγματεύονται 35 κεφάλαια, όταν μετά πρέπει να μεταγράψουν το ενωσιακό δίκαιο, χρειάζεται να εφαρμόσουν μόνο 20 κεφάλαια και χρειάστηκε τελικά να ασχοληθούμε με νομοθεσία που δεν ίσχυε πια. Δεν νομίζω ότι ε, ενημερώθηκαν καλά τα κείμενα μετά την μεγάλη διεύρυνση. Και το τρίτο, Είχαμε Δανούς, Ολλανδούς και Βρετανούς να κάνουν γύρω των πρωτευουσών και να λένε Ευρώπη μόνο εκεί που χρειάζεται. Πώς ε, έχετε αντιληφθεί αυτό το μήνυμα και πώς το εφαρμίζετε. Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Μου ήρθε βέβαια η ιδέα να ζητήσω από τον κύριο Τίμερμανς να παραλάβει ε, αυτά που είπε για το πώς αντιμετωπίστηκε από τη Γερμανία η Πορτογαλία. Θέλω όμως καλύτερα να θέσω μία ερώτηση για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών κρατών και επενδυτών. Ε, επενδυτών και κρατών ξέρω ότι θα γίνουν περαιτέρω επαφές για να βελτιώσουμε την κατάσταση για το θέμα αυτό, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν και κατά πόσο θα συμπεριληφθεί αυτός ο μηχανισμός ISDS στη συμφωνία TTIP. Αυτές οι βελτιώσεις ε, θα έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ε, υιοθέτηση ρυθμιστικών ε, διατάξεων για το πώς θα λειτουργούν αυτά τα διαιτητικά δικαστήρια και με άλλους μηχανισμούς και δυνατότητα προσφυγής μάλιστα κατά των αποφάσεων αυτού του μηχανισμού με στόχο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα περιοριστεί η δικαιοδοσία των ε, κρατών των, ε, συγγνώμη, των δικαστηρίων των κρατών μελών σε περιπτώσεις ε, διαφορών. Ούτως ή άλλως οποιοδήποτε μηχανισμός διαιτησίας δεν μπορεί να περιορίζει τη δικαστική εξουσία ενός κράτους. Προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά. Διότι συνήθω είναι εναλλακτική μέθοδο επίλυση διαφορών η διαιτησία. Εναλλακτική, διαφορετική από τι δικαστικέ αρμοδιότητε. Θα εξακολουθήσει να είναι εναλλακτική ή πάντα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης των αποφάσεων αυτών των ε, διαιτητικών δικαστηρίων. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το σύστημα ISDS και να μην ε, οδηγήσει σε περιορισμό των εθνικών δικαιοδοσιών. Μήπως μετά μας πείτε τίποτα για όλα αυτά. Σαλ Γκέρνς. Ευχαριστώ. Μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Τίμερμαντς. Θα θυμάστε την απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από μερικού μήνε να ορίσει τον κύριο Στυλιανίδη συντονιστή τη Ένωση για την αντιμετώπιση του έμπολα. Η απόφαση αυτή είναι σωστή. Μπορεί, αλλά ο τρόπος λήψης της ήταν προβληματικός. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει ένας επίτροπος θα αναλάβει το συντονισμό της αντιμετώπισης του έμπολα. Νομίζω ότι οι συνθήκες ε, περιέχουν επαρκή βάση για να παίρνει η Κομισιόν τέτοιες αποφάσεις χωρίς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η απόφαση θα μπορούσε να έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορούμε να αναφέρουμε για το Συμβούλιο είναι ότι ακόμη δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε επιβεβαιωθεί βέβαια από το, δικαστή, από το Κοινοβούλιο, αλλά δεν είχε ακόμη αναλάβει τις αρμοδιότητες της. Μπορείτε να μας ε, σχολιάσετε αυτή την απόφαση. Αυτά. I think there was a question on... Σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα της Γερμανίας, ε, πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, φορολογήσει για τη χρήση των ε, οδικών υποδομών, αλλά δεν θα πρέπει να υφίστανται αντικές διακρίσεις των, για τους πολίτες δεν είναι δυνατόν να υφίστανται διόδια τα οποία να παραβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία Δηλαδή, ε, αν κάποιος ε, οδηγήσει μέχρι την Γαλλία, χρειάζεται να πληρώσει για τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου. Όλοι πληρώνουν, και οι Γάλλοι πολίτες. Ε, αυτή την έννοια δεν γίνεται διακριτική μεταχείριση. Το θέμα δεν είναι αν μπορεί να εισάγει κανείς διόδια, αλλά για το κατά πόσον μπορεί αυτό να περιοριστεί για συγκεκριμένου ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά τον, ε, το ελάχιστο, τον ελάχιστο μισθό, δεν απαγορεύεται από την, Ευρωπαϊκή, από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία έχει αυτό το, αυτή τη μέθοδο και δεν είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να προσβληθούν, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί με τον αλφίτο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για την δημόσια, δημόσιο διάλογο, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά. Μερικές φορές σε διάφορους ευρωπαϊκούς κύκλους βλέπω ότι ορισμένοι αμυντικά ε, λένε τόσο πολλά κάνουμε για την Ευρώπη γιατί δεν μας ευγνωμονούν. Ε, δεν είναι πολύ καλό αυτό, δεν βοηθάει. Θα πρέπει ε, να παρουσιάσουμε το έργο μας στους Ευρωπαίους πολίτες μέσα στο πλαίσιο ενός ανοιχτού πολιτικού διαλόγου και αυτό πιστεύω θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ως ακαδημαϊκός ε, καθηγητής πανεπιστήμιο ε, ερχόμουν σε επαφή με διάφορους ανθρώπους που θεωρούσαν ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να ε, ταξιδεύουν και να εργάζονται να φοιτούν σε άλλα κράτη-μέλη. Και του εξηγούσα ότι τώρα μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό, αλλά όταν ήμουν εγώ μικρό και νέο δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό. Οπότε η, τα ωφέλη τη Ενωμένη ΕΕ Ευρώπης ε, έχουν ενταχθεί τόσο πολύ στην καθημερινή ζωή που τίνουμε ε, να τα γνούμε, να μην τα βλέπουμε και ε, αυτό είναι ένας κίνδυνος. Μερικές φορές μιλώ εγώ στα εγγόνια μου για τα... Ε, ε, στα παιδιά μου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταστραφεί. Ότι είναι μόνιμο. Δεν ισχύει αυτό. Ε, εγώ είχα δουλέψει στη δεκαετία του 90 ως νέος διπλωμάτης στη Βαλτική και εκεί KGB σκότωνε διάφορους ανθρώπους γιατί προσπαθούσε να, τηρήσει, να διατηρήσει ε, την, ε, τις χώρες της Βαλτικής ε, στην Σοβιετική Ένωση και τώρα έχουμε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρα της Βαλτικής και ήθελα να πάρω τα παιδιά μου να τα πάω εκεί για να τους δείξω αυτή την περιοχή και να συγκρίνω τη δική τους εμπειρία με τη δική μου. Η δική μου δεν είναι και τόσο παλιά, 30-35 χρόνια πριν. Σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να εστιάσουμε τη συζήτηση στην Ευρώπη. Αν δείτε ε, τους ανθρώπους στο Μαϊντάν, στο Κίεβο, ε, βγαίνουν στους δρόμους με ε, σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Ε, γιατί για αυτούς η σημαία αντικατοπτρίζει αξίες. Δεν είναι επειδή υποστηρίζουν την Κομισιόν, το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Εμείς αυτές τις αρχές τις θεωρούμε σαν κάτι δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο. Αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνει για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και όλοι πρέπει να συμμετάσχουν. Γιατί πολλοί, όλοι πιστεύουμε ενδεχομένω ε, τις ίδιες αξίες, αλλά δεν συμφωνούμε όλοι για το πώς θα πρέπει να είναι η θεσμική διάρθρωση, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και σε αυτό η Κομισιόν θέλει να συμμετάσχει. Καλύτερη νομοθεσία. Ναι. Δεν σημαίνει λιγότερη νομοθεσία. Ελπίζω να σημαίνει και αυτό, αλλά όχι απαραίτητα. Καλύτερη νομοθεσία σημαίνει νομοθεσία που υπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 5-6 χρόνια, μέχρι πριν από 5-6 χρόνια, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πίστευαν ότι η Ευρώπη τους ωφελεί. Μπορώ να πω σήμερα ότι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι βαρύδι δεν τους βοηθάει να αυξήσουν τις προσλήψεις. Ε, εγώ θα κρίνω την επιτυχία μου από το κατά πόσον στο τέλος της θητείας μου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λένε ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους επιτρέπει να μειώσουν τη γραφειοκρατία, τη γραφειοκρατία τους επιτρέπει να κάνουν περισσότερες προσλήψεις και τους επιτρέπει να δουλεύουν πιο ελεύθερα χωρίς να μειώσουμε, χωρίς να κατεβάσουμε τον πύχη των ε, ε, κοινωνικών παροχών και διευκολύνσεων. Δεν είναι εύκολο, αλλά και ποιος θέλει το εύκολο, ποιος κυνηγάει το εύκολο. Επίσης, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και μια θετική ατζέντα για τα εθνικά κοινοβούλια, χωρίς όμως να πέσουμε στην παγίδα να δώσουμε στα εθνικά κοινοβούλια το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Κάποια κοινοβούλια το θέλουν αυτό. Όχι. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνεισφέρουν χωρίς όμως να τους δώσουμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Γιατί κάτι τέτοιο θα παρέβαινε και τη συνθήκη. Θα πρέπει έτσι κι άλλως να την αλλάξουμε και βέβαια μπορεί να την αλλάξουμε, αλλά δεν είναι και το θέμα. Θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο πολιτικό τρόπο να συμπεριλάβουμε και τα εθνικά κοινοβούλια. Χωρίς να χρειαστεί αλλαγή συνθήκης. Τώρα, για τις εκλογές στην Ελλάδα. Εγώ έχω εκλεγεί έξι φορές το Εθνικό μου Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να κάποιος της Βρυξέλλης κάθε φορά να έλεγε ε, κάτι δύο μέρες πριν τις εκλογές για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι δύο <laughs> μέρες και ε, οι ελάχιστες εν πάση περιπτώσει μέρες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα δεν θα τολμήσω να πω τίποτα. Ε, θα μπορούσα να πω κάτι διπλωματικό ε, αλλά επειδή σας σέβομαι θα σας πω ότι δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σας γιατί ξέρω ότι οτιδήποτε και να πω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τον α ή τον β τρόπο. Ε, αν θέλετε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα μετά τις εκλογές θα είμαι στη διάθεσή σας. Η σύνθεση των επιτροπών είναι κάτι που έχει σχέση με το δικό σας κοινοβούλιο, όχι με την Επιτροπή, όχι με την Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν μπορεί να αποφασίσει πώς εσείς ε, συστήνετε τις Επιτροπές σας. Αν δεν κατάλαβα καλά, παρακαλώ ε, διορθώστε με, αλλά έτσι κατάλαβα την ερώτησή σας. Δυστυχώς χωρίς ε, μικρόφωνο μιλτής. Yeah, yeah, uh, sir, I, I understand that point perfectly well. Ε, Κατάλαβα τι λέτε. Απόλυτα. Αλλά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την επιτροπή, μάλλον ε, ποια θα είναι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την επιτροπή, είναι απόφαση την οποία λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι καταλαβαίνω χρησιμοποιεί τον κανόνα του DONT, ε, που χρησιμοποιείται και αλλού. Η μόνη φιλική συμβουλή που μπορώ να δώσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είναι δική μου, δικό μου πεδίο, ε, είναι ότι σύμφωνα με τη δική μας Ολλανδική εμπειρία όταν ε, έχουμε πολυκομματική βουλή ε, γίνονται πιο, δυσ, γίνεται πιο δυσχερής η χρήση του κανόνα DON'T. Τώρα βέβαια αυτό είναι τελείως φιλική συμβουλή. Τώρα, Ο κύριος Καστάλτο ξανά. Thank you. Uh, it was just... Θέλω να διευκρινίσω. Να σας πω δηλαδή ότι δεν ρωτούσα την Κομισιόν να τροποποιήσει τους κανόνες του Κοινοβουλίου. Και να αλλάξει η Κομισιόν τον κανόνα don't. Απλώς σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις να αυξήσει τον αριθμό των εδρών. Ούτε ώστε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες να παίξουμε. Γιατί όταν έχουμε μόνο πέντε θέσεις σε μία επιτροπή, ας πούμε, σε, σε μία ομάδα, κάποια πολιτική ομάδα αναγκαστικά θα αποκλειστεί. Γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση. Τι να σας πω. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Και μια και εγώ είμαι από την πολιτική σας ομάδα, το να ζητήσω περισσότερη γραφειοκρατία δεν νομίζω ότι είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν περίμενα από εσά να ζητάτε περισσότερη γραφειοκρατία. Όταν υπάρχουν περισσότερα πολιτικά κόμματα στην Ολλανδία, ξέρω ότι τα μικρά θέλουν να γίνει οτιδήποτε, ούτως ώστε να ακούγονται οι περισσότερες, περισσότερες απόψεις, περισσότερες φωνές. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που θέτεται. Ευχαριστώ κύριε Πλένκοβιτς που μιλήσατε για το θέμα της μετάφρασης. Θα το έχω υπόψη μου στο μέλλον. Επίσης να ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της Επιτροπής δεν προβλέπουμε να γίνει νέα διεύρυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τη διεύρυνση, τη διαδικασία διευρύνσεων. Ε, υπάρχουν πράγματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και έχουμε τεράστιες ευθύνε για να συνεχίσουμε τη διαδικασία διευρύνσεων. Αλλά αν μου λέτε, αν είναι δανέζικη, ολλανδική ή βρετανική, ας πούμε, η ατζέντα, σας παραπέμπω στις δημόσιες δηλώσεις του Σούλτ, του Ιούνκερ, του Φερχόφστατ και όλων των ηγετών. Όλοι είπαν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι μεγάλη για τα μεγάλα και μικρή για τα μικρά. Θα πρέπει να ξαναδούμε τις προσπάθειές μας. Τα υποσχέθηκαν αυτά προεκλογικά. Και θα πρέπει να το κάνουν μετεκλογικά. για το πρόγραμμα της ε, Κομισιόν, για το ReFeed, για την καλύτερη νομοθεσία, για την επιθυμία που έχουμε για να συμφωνήσουμε ε, σε μια διαθεσμική βάση για μια καλύτερη νομοθεσία. Για όλα αυτά και τα τρία θεσμικά όργανα εμπλέκονται. Για το SDS, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτών Κρατών. Να πω το εξής, ότι σε διμέρες επίπεδο υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι μηχανισμοί μεταξύ των κρατών μελών. Μετα... Μερικές φορές ε, θεωρείται ο διάβολος που θα θέσει τέρμα στη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Γιατί εντάξει έχουμε εμπειρία από αυτό το μηχανισμό. Αλλά πόρα απέχουμε από την επίτευξη μιας τέτοια συμφωνίας. και πολύ μακριά είμαστε από ένα TTIP. Έχω την αίσθηση ότι τα δικαιώματα των πολιτών, εάν δεν ε, αντιμετωπίζονται σωστά, εγώ θα πω όχι στο ISDS. Και θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός ως προς αυτό. Αν μου με ρωτάτε σήμερα, να σας πω τι λέμε όταν εννοούμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι δεν θα περιορίσουμε την πρόσβαση στην, των Ευρωπαίων πολιτών στην εθνική νομοθεσία. Ε, έχω να σας πω ότι η αρχή ισχύει και εμείς θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε αυτή την αρχή. Θα τη βάλουμε αυτή την αρχή, θα την ενσωματώσουμε σε ένα ISDS και θα ήταν πολύ χρήσιμη και για ένα TTIP. Εάν αυτή η ιδέα δεν υπάρχει, ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε ολόκληρη την, ολόκληρο το μηχανισμό. Δεν, είμαι, δεν έχω αιμονές για το ISDS, αλλά δεν απορρίπτω οποιονδήποτε μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Γιατί μερικές φορές τέτοιοι, μηχανισμοί έχουν εξυπηρετήσει πολύ τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους πολίτες. Για το ποιος θα είναι υπεύθυνο για την κρίση του έμπολα, στην αρχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαμε δύο επιλογές. Είτε η Κομισιόν να είναι υπεύθυνη, είτε να υπάρχει ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας, οποιοδήποτε, που θα είναι εξάρτητος ή από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παίξουν αυτό το ρόλο. Τελικά είπαμε ότι θα κρατήσει η Κομισιόν την ευθύνη και Ποιο θα είναι ο υπεύθυνο, ο Επίτροπο Τηλιανίδη. Αυτό κάναμε. Έκανε θαυμάσια δουλειά. Ταξιδεύει με μεγάλη ενεργητικότητα. Ναι, η Κομισιόν θα μπορούσε να έχει αποφασίσει μόνη τη ότι ο Χρήστο θα έπαιζε αυτό το ρόλο. Αλλά πριν ληφθεί αυτή η απόφαση, έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τις σχέσεις, ας πούμε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κομισιόν. Δηλαδή, αν θα ήταν κάποιο από την Κομισιόν, θα ήταν κάποιο εξωτερικό. Νομίζω ότι τα απάντησα όλα τα θέματα. μισή μήνες ήσασταν στην Κομισιόν. Ε, πώς αισθάνεστε? Όλα καλά? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν σας ελέγχω, δεν σας λέω τίποτα. Μόνο δυόμιση μήνες πέρασαν. Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι το να έχουμε ένα τακτικό διάλογο με τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές βοηθάει γιατί ξεκαθαρίζονται ιδέες και κρατάμε το κοινοβούλιο ενήμερο για το τι κάνει η Κομισιόν. Μ' αρέσει κάτι τέτοιο. Θέλω να συνεχιστεί. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Εάν όλοι συμφωνήσουν ότι πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Α, μάλλον συμφωνούμε όλοι με αυτή την ιδέα ότι πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά πάντα θέλουμε να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία των άλλων, όχι τη δική μα. Έτσι. Και θέλω να το λαμβάνω αυτό υπόψη μου όταν κάνω τι προτάσει μου. Να λαμβάνω υπόψη και τη δική μου γραφειοκρατία. Σα ευχαριστώ όλοι, κύριε Χιούμπνε, και καλή τύχη για τη συνέχεια.